Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ε, καθίστε όμως, παρακαλώ. Ε, αφήστε ήσυχους τους βουλευτές, παρακαλώ. Σημείο 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. το σημείο 9 κατευθυντήρε γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εντολή του ειδικού απεσταλμένου για την πρόωση τη θρησκευτική ελευθερία αναβάλλεται κατόπιν αιτήματο ε, του εισηγητή σε μια επόμενη συνεδρίαση. Αν ε, δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, η μερίσια διάταξη εγκρίνεται με αυτήν την αλλαγή. Σημείο 2 δεν έχω ανακοινώσεις να κάνω. Σημείο 3 πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 10 Ιουλίου, της 3ης Σεπτεμβρίου και της 27ης Σεπτεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά εγκρίνονται. Μετά περνάμε στην ψηφοφορία. Όπως ξέρετε, είναι μακροσχελέστατη. οπότε ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Η πρώτη ψηφοφορία αφορά την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ΚΕΠΑ. Ο εισηγητής έκανε εξαιρετική δουλειά. Είναι τόσο εξαιρετική που δεν χρειάζεται να λάβει τον λόγο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσω την ψηφοφορία εάν συμφωνείτε. Πού είναι ο κατάλογος. Μάλιστα. Ξεκινάμε. Συμβιβαστική 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές θα την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 52 ψήφισαν. Απορρίπτεται. 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ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 Προφορική τροπολογία. Ναι, κύριε Ποστινάρου. Κύριε Πρόεδρε, θα είχατε την καλοσύνη να ξεκαθαρίσετε πόσα το... τέσσερις βουλευτές χρειάζονται μάλιστα για να φέρουν κάποια αντίρρηση. Κοιτάξτε, η προφορική τροπολογία έχει στόχο να επαναφέρει τα θέματα αυτά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και λέει παραβιάζει τις ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ιεμένη και τις αδιάκριτες επιθέσεις κατά μάχων από την Σαουδαραβική Συμμαχία. Ζητάει άμεση κατάπαυση του πυρός ε, και να επαναληφθεί ο διάλογος υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και να υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και επιμένει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση δεν αναφέρεται πουθενά η, η εμένη. Και νομίζω ότι είναι η σημαντικότερη κρίση που υπάρχει σήμερα. Ωραία, σας ευχαριστώ για την προφορική τροπολογία. Τέσσερις συνάδελφοι πρέπει να είναι κατά. Πόσοι υπάρχουν. υπάρχουν. δύο, 3, τέσσερις, πέντε, έξι.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 αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 καταπίπτει, 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθηκε άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 38 υπέρ 7 ψήφι κατά 11 αποχές. Κυρία Λέζινγκ, παρακαλώ. Έχουμε υποβάλει μια έκθεση τη σημειοψηφίας και την έχουμε ήδη αποστείλει στην γραμματεία. Σας ευχαριστώ και το περίμενα. Γεια σου Τζούλιαν. Λοιπόν, Αχ, όχι, ε, σημείο 5. Ανησυχίε ω προ τον σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεξαγωγή επιχειρήσεων από ιδιωτικέ στρατιωτικέ εταιρείε. Ο κύριο Κάρσκι θέλει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια για ένα σημαντικό θέμα που το εξετάζει η ΟΗΕ. Πρόκειται για καταστάσεις στις οποίες έχουμε ιδιωτικέ ε, στρατιωτικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν δράση εξ ονόματος κρατών ή ακόμη και ιδιωτικέ εταιρείε οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διεθνείς ε, συγκρούσεις και με αυτόν τον τρόπο είναι δύσκολο να αποδώσει κανείς ευθύνες. σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπινών δικαιωμάτων και αυτό δημιουργεί προβλήματα με την λογοδοσία. Το φαινόμενο γίνεται όλο και πιο συχνό έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες ιδιωτικέ εταιρείε να δραστηριοποιούνται σε στρατιωτικέ επιχειρήσεις και με βαρύ οπλισμό. Παρά το γεγονό ότι υπάρχει ήπια ρύθμιση soft law, ε, δεν είναι ικανοποιητικό το διεθνές ε, ε, πλαίσιο για αυτές τις εταιρείες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία έχει ξεκινήσει από την Επιτροπή Ντροά και διευκρινίζω ότι μιλούμε για εταιρείε οι οποίε δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία που είχαμε. Καταλήξαμε στις συμβιβαστικέ τροπολογίες για όλα τα θέματα και σας ζητώ να υποστηρίξετε την έκθεση. Σας ευχαριστούμε που μας παρουσιάσατε την έκθεσή σας και σε τι αναφέρεται, οπότε ξεκινάμε με τις τροπολογίες. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για τη συμβαστική τροπολογία 9 λοιπόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε την τροπολογία 145 ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα την ελέγξουμε την 149. Καλώς, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεν ψηφίσουμε για την 158. Περνάμε στη συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την τροπολογία 165 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 166. Τμηματική ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 166. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μικρή διαφορά. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α ελέγξουμε την 167. Θα τραβήξει πολύ ψηφοφορία νομίζω σήμερα. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 179 κύριος Μπούχνερ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 181 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 185 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 186 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 187. Πέρας. Απορρίπτεται. 189 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 191 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 191 ηλεκτρονικά. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπούχνερ. Περνάμε στη συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε τη συμβαστική τροπολογία 15, άρχη τη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 202. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. «204 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 205 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 208 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 209 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 210 υπέρ, κατά, Αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 217 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά απόχέ. να ελέγξουμε τη... 218 λέει ο Πρόεδρος. Πέρας. Εκρίνεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 224 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 224. άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 225 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε και τη 225 Εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε στην συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20, συμβαστική 21 υπέρ Ζητώ συγγνώμη. 162 υπέρ, κατά, αποχές. Θα πρέπει να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά, την 162. Πέρας. Απορρίπτεται. 237 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 238 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 238. Απορρίπτεται. 240 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 241 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 242 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 243 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 245 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 246 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 246 ηλεκτρονικά αρχή τη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 247 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 248 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 249 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 224 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, να ελέγξουμε, να ελέγξουμε την τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τρία τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, θα πρέπει να ελέγξουμε τη συμβαστική τροπολογία 3. Πέρας, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33. Να ελέγξουμε την 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ας εστιάσουμε πραγματικά στις ηλεκτρονικούς ελέγχους εκεί που χρειάζεται. 33 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37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 θα πρέπει να ελέγξουμε την τροπολογία 43 και 44. άρχιτη η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για τις 46. Πάμε στις 48 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αλλά ας την ελέγξουμε. 46 λοιπόν. Πέρας. Απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα την ελέγξουμε τη 47. Καλώς άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 48 και 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. 48. Πέρας. Εγκρίνεται. 50, 51, 52 και 53 υπέρ. Κατά. Άποσες, Ελέγχουμε και αυτές. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 54, πάμε 55 και 56 υπέρ, κατά, άποχες. Να την ελέγξουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 58, 59 και 60 υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε και αυτή ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με σαφή πλειοψηφία. Έλαβαν χώρα συνεδριάσει με τους κοιότητες συζητητές για να βρεθούν κάποιοι συμβασμοί. 63-66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. να ξαναρωτήσω, έλαβαν χώρα στι συναντήσει με τους κοιόδη συζητητέ του, ώστε να υπάρξουν κάποιοι συμβιβασμοί σε σχέση με αυτή την έκθεση. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Πάμε στι 68, 69, 70 και 71. Υπέρ, κατά, απόχε. Θα πρέπει να ελέγξουμε και αυτέ τι τροπολογίε ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνονται. 73 υπέρ, κατά, αποχές. Εδώ, συνάδελφοι, δεν τους βλέπω να σηκώνουν τα χέρια, οπότε θα πρέπει να την ελέγξουμε και αυτή την τροπολογία ηλεκτρονικά. Πάντα για την τροπολογία 73. Πέραση της φοφορίας. Εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75 και 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80, 81 και 82 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε αυτές τις τροπολογίες. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 και 87 υπέρ. Κατά. Αποχές Ας ελέγξουμε. Τις 86 και 87. Απορρίπτονται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, το 89 υπέρ,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 100 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την τροπολογία 100. Πέρας. Απορρίπτεται με σαφή πλειοψηφία. 101 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102 τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 102 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την ε, τοπολογία 105 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγξουμε και την 106. εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 108 έως 110 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και άλλη συμβαστική τροπολογία, τι θαύμα. Περ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 125. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται 125, 126 τώρα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται 127 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται 128 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχέ. Ελέγχουμε τροπολογία 2.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 συνάδελφος δεν έχει ψηφίσει ακόμα. Ξυπνήστε, καλός πέρας. Απορρίπτεται λοιπόν το σύνολο της έκθεσης. 34 ψήφοι κατά και 25 υπέρ. Thank Σας ευχαριστώ. Συνεχίσουμε με το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής είπατε εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής, για θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πρέντα. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η ομάδα μου δεν συμφωνεί με το γεγονός ότι γίνονται αναφορές σε κρατη σε αυτή την έκθεση, γιατί δεν το θεωρούμε σωστό. Δεν το θεωρούμε καθόλου σωστό. Ήθελα να το διευκρινίσω, να το επισημάνω. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέντα για αυτήν την παρατήρηση. Ο εισηγητής μήπως θα ήθελε το λόγο. Ελάτε. κύριο Χάν. Θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω μια ανησυχία μου. Μιας και το ΕΛΚ διατυπώνει αυτή την ένσταση αν θέλετε. Όσο δεν το παρακολουθείτε, το ζήτημα είναι το ζήτημα η ελευθερία, η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της έκφρασης σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την έκθεση για να, την, για να προασπίσουμε την ακαδημαϊκή ελευθερία σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί κακό προηγούμενο εάν θεωρήσουμε ότι είναι απαράδεκτε τροπολογίε οι οποίε αναφέρονται σε κράτο μέλο τη Ένωση. Έχουμε μια παγκόσμια στρατηγική για την, τα ανθρώπινα δικαιώματα και λέμε ότι η εξωτερική και η εσωτερική διάσταση θα πρέπει να είναι συνεκτικέ μεταξύ του. Πιστεύω ότι αν δεχτούμε αυτή τη φιλοσοφία η θα είναι σαν όπιστο χωρούμε, κατά την άποψή μου. Σα ευχαριστούμε κύριε Χάν. Θα ήθελε κάποιο άλλο το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Συνάδελφοι, να εξηγήσω λίγο τι γίνεται, λέει ο πρόεδρος. Τι συμβαίνει. Έχω λάβει ενστάσεις όσον αφορά το παραδεκτόρισμα ανθρωπολογιών. Με email από συνάδελφο από το ΕΛΚ, και έχω επίση και την απάντηση του εισηγητή. Γνωρίζετε ότι αποτελεί αρμοδιότητα του Προέδρου να αποφανθεί επί της κατά πόσο μια τροπολογία είναι αποδεκτή. Συμβουλεύτηκα τη γραμματεία και εξέτασα βεβαίως μόνο εκείνα τις τροπολογίες για τι οποίες υπευλήθη επίσημα αίτημα. Στη, στην Σύνοδο των Προέδρων έχουμε συμφωνήσει να γίνεται πλήρες συμβασμός των αρμοδιοτήτων κάθε επιτροπής και της Επιτροπής ΑΦΕΤ στην περίπτωση αυτής της έκθεσης που, για την οποία θα ψηφίσουμε. Έχουν υποβληθεί διάφορες τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στο ιστορικό πλαίσιο ή γενικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρουν γενικά μιλώντας ότι ε, επιθέσεις κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας μπορούν να συμβούν και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θεωρώ ότι είναι αποδεκτές, παραδεκτές, γιατί και ως εκ τούτου απορρίπτω το αίτημα της κυρίας Μπέξελ για την τροπολογία 4. Υπάρχουν όμως και ένα άλλο σύνολο τροπολογιών που αναφέρονται για, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητούν ανάληψη δράσης και αυτές τις θεώρησα μη παραδεκτές. Εμείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ΑΦΕΤ θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση σε σχέση με την εξωτερική διάσταση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοια ζητήματα αποτελούν αρμοδιότητα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Αυτή είναι η απόφαση του Προέδρου. Εάν σα ικανοποιεί, μπορείτε να μου το πείτε. Αν όχι, μπορείτε να καταγορήσετε τη γραμματεία. Αστείευεται ο Πρόεδρο. Προσπάθησα να ε, λάβω μια απόφαση την οποία να μπορούν να δεχτούν όλοι οι συνάδελφοι με βάση του κανόνε. Εάν δεν θέλει κάποιο άλλο συνάδελφο το λόγο, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε, έτσι για να ζεσταθούμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα ψηφοφορίας. Ξεκάθαρα εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβα... 64 υπέρ κατά εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ για την 67 του κ. Μπούχνερ. της ψηφορίας. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 69 θεωρήθηκε μη παραδεκτή. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνε. απορρίπτεται. 72 υπέρ, κατά, Αποχέ. Α ελέγξουμε την 72, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, Αποχέ. απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε ψηφίστε για την 90 παρακαλώ. Πέρας ψηφορίας εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές Μάλλον απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. απουσίε. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. απουσίε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. απουσίε. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. απουσίε. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. απουσίε. Εγκρίνεται. Ιδεολογικέ σκέψει 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές μου φαίνεται ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε ψηφίστε παρακαλώ για την 20. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ε, Α ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ για την συμβαστική 12. Πέρας ψηφορίας εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε, ψηφίστε για την 30 παρακαλώ. Πέρασε τις φορές. Εγκρίνεται. Συμβασική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγξ, ας ελέγξουμε, ψηφίστηκε 34. τη εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 όχι. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ψηφίστε για τη 40 παρακαλώ. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. Ξεκάθαρα. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε ψηφίστε για τη 42. Πέρας φορές. εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές. Ε, απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές. Ε, απορρίπτεται.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 και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την έκθεση όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίστε παρακαλώ. Άλλος ένας συνάδελφος πρέπει να ψηφίσει. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται 56, με 56 ψήφους υπέρ συγχαρητήρια στην εισηγητή. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο Συμφωνία υπό 7. Συμφωνία υπομορφή ανταλλαγή επιστολών μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Βασιλείου του Μαρόκου για τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθμών 1 και 4 τη Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Βασιλείου του Μαρόκου. Ο κύριο Βίστισεν είναι ο εισηγητή. Θέλετε τον λόγο, όχι. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο της γνωμοδότησης άρχεται η ψηφοφορία τρεις συνάδελφοι δεν έχουν ακόμα ψηφίσει πέρας εγκρίθηκε 44 υπέρ 17 κατά Περνάμε. Ποιο είναι αυτό. 8. Ίδιο μου φαίνεται. Α, είναι το ψήφισμα που το συνοδεύει. Ωραιότατα. Έχουμε κατάλογο ψηφοφορίας. Α, Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18 ε, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε ποιος είναι υπέρ άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. να σαφής πλειοψηφία. Φρόιντ υπέρ. Κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 39 Πέρασε. απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε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 να την επαληθεύσουμε, αρχή η ψηφοφορία. Πέρασε. Έχει εγκριθεί 65 υπέρ, κατά αποχές, το 66 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 67 υπέρ. Να ελέγξουμε το 66, ωραία, υπέρ του κυρίου 5. Πέρας, εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές να την επαληθεύσουμε. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83, την ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του τη ψηφοφορία. Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Πολύ αργά. Πέρασε. Συγχαρητήρια στον Αντιπρόεδρο. Το θέμα 9 έχει αναβληθεί όπως σας είπα. Περνάμε στο σημείο 10 θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού στον τομέα τη πυρηνική ασφάλεια, του μηχανισμού Μηχανισμό Γειτονία Ανάπτυξη και Διεθνού Συνεργασία βάσει τη συνθήκη Ευρατόμ. Εισηγητή είναι ο κύριο Αυστρεβιτσίου. Θέλετε τον λόγο. Όχι. Οπότε προχωράμε. Συμβαστική ένα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δύο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 αποσύρεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 ψηφίζουμε. Υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σε συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 46 αντρική 1 υπέρ, κατά αποχές να την επαληθεύσουμε αρχιτή ψηφοφορία. Δεν έχουν ψηφίσει όλοι οι συνάδελφοι. Πέρας. Ε, σαφώς. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές θα την επαληθεύσουμε αρκετή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Υπέρ κατά αποχές 13 ε, υπέρ κατά αποχές 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ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 κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε, Εγκρίθηκε με 51 ψήφου υπέρ κατά. Σημείο 11. Δικέ διατάξει ότι έχουν το στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, ο οποίο υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και του Μηχανισμού Εξωτερική Χρηματοδότηση. Ε, Καστάλτο, θέλετε τον λόγο, όχι, δεν είναι εδώ. Θα ήθελα να σας ε, ε, υπενθυμίσω συνάδελφε ότι με βάση το άρθρο 53 παράγραφος 2 του ε, καταστατικού ε, προβλέπει ότι οι εκθέσεις μας θα πρέπει πάντοτε να αφορούν στον τομέα αρμοδιότητας αυτής της Επιτροπής ε, και κατά συνέπεια αποφάσισα ότι εξή τροπολογίες δεν είναι παραδεκτές 68, 72, 87 και μία ακόμα του κυρίου Χάνοκ Αυτές οι τέσσερις λοιπόν τροπολογίες δεν θα ψηφιστούν και περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκατέσσερα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15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 απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εδώ τώρα έχουμε ε, ψηφοφορία και τις 77 ως 82 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Και πάλι το ίδιο, 23 ως 26 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για τις 23-26. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ, είμαστε εν μέσω ψηφοφορίας. Δεν μπορείτε να συζητήσετε τόσο τη αίθουσα. Πέρα τη ψηφοφορίας απορρίπτονται. 27 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ και 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 89 λοιπόν, ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται εγκρίνεται 91 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε τροπολογία 91, αρχή ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε την 97. Απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε την 99 άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 107, δεν είναι παραδεκτή, 108 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ, κατά αποχές. Θα ελέγξουμε την 109 ηλεκτρονικά αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 110. Κύριο Σπάιτ. Έχει υποβάλει πολλές τροπολογίες. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές,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 121 κύριο Στάνοκ υπέρ κατά αποχές εκρίνεται. Έχουμε ψηφοφορία για τις 123, 125, 127, 129, 131, 132, 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Και πάλι συνολική για 122, 124, 126, 128, 130, 132 υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά αυτές τις τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 135 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά. Τηλογικές σκέψεις. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Κύριος Καστάλλου Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45. Υπέρ κατά... Α, όχι. Κατά πίπτη. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Με τον κύριο Πίτσολα όμως τώρα. 52 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε τροπολογία 5, άρχη της ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε την 56 ηλεκτρονικά. Πέρας απορρίπτονται με σαφή πλειοψηφία 57 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτονται 6 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 59 καταπίπτει 10 υπέρ κατά αποχέ. θα ελέγξουμε την τροπολογία 10 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Με μικρή διαφορά απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν τώρα στο στην ηλεκτρονική ψηφοφορία από του συνόλου του σχεδίου γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέσσερι συνάδελφοι δεν έχουν ακόμα ψηφίσει. Πέρας τη ψηφοφορία. 47 ψήφοι υπέρ, 4 κατά. Συγχαρητήρια. Και περνάμε τώρα στο σημείο 12 της Μέσης Διάταξης, Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Ιαπωνίας αφετέρου. Εισαγητής είναι ο κύριος Πέτερλε. Θέλετε το λόγο? Αυτή την όμορφη και τη μέρα, ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας για μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας που να είναι τόσο πλήρης και στρατηγικής σημασίας. Έχουμε δύο παράλληλες διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε δύο συμφωνίες εταιρική σχέσης και στρατηγικής σχέσης, η και SPA. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και επίσης τον πρέσβη της Ιαπωνίας, για την ε, πολύ καλή συνεργασία που είχαμε επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πέτερλε. Μήπως θα ήθελε κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Επομένως, θα ξεκινήσουμε ε, για το προσχέδιο σύστασης που πρέπει να ψηφιστεί ηλεκτρονικά με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε φορές. Εγκρίνεται με 47 ψήφους υπέρ και 2 κοτά. Και τώρα ερχόμαστε στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 81 τροπολογίε είχαν υποβληθεί. Έχουμε 14 συμβαστικέ από τον εισηγητή, ο κύριο Πέτερ Λεπάντα. Α ξεκινήσουμε. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά εγκρίνεται, 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 34 κύριε, του κ. Μάρτιν υπέρ κατά αποχές. Να σε ελέγξουμε, ψηφίστε για την 34 παρακαλώ.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 αντικαθιστούμε τη λέξη deplores with, με τη λέξη regrets. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ψηφίστε για την 74. Πέρας ψηφορία. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ψηφίστε για την 75 παρακαλώ. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, Δεν βλέπω μεγάλη συμμετοχή από τους συναδέλφου. οπότε θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. στι ψηφορίας. Εγκρίνεται. Πολύ. 77 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ε, απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ο κύριο Πέλτερ 4 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχέ. Απορρι... Εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχέ. Εγκρι... Απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Παραπομπές 1 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 3. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρες ψηφοφορίας απορρίπτεται η 3. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας φορείες, με 43 ψήφους υπέρ, 2 κατά, εγκρίνεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία, τη ψηφοφορία και μάλιστα πέντε λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα. Επομένω, δικαιούμαστε ένα διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε στι 10.30. So. So, ladies and gentlemen, please be seated. Let's... continue. Κυρίες και κύριοι, καθίστε να συνεχίσουμε την συνεδρίαση. Επειδή ήμασταν πολύ γρήγοροι στις ε, ψηφοφορίες, έχουμε προχωρήσει λίγο στην ημερήσια διάταξη. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ξεκινήσουμε τώρα το θέμα 14. Θέσμιση του, θέσπιση του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας. Συνάδελφοι, στο επόμενο ΔΕΛΤΑΠΗ 2021-2027 ο μηχανισμός Προταξιακής βοήθειας θα συνεχίσει να στηρίζει χώρες υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες. Συγητές είναι ο Χωσέ Ιγνάσιο Σαλαφράνκα και ο κύριος Φλέκενστάιν από τους σοσιαλδημοκράτες. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Κύριε Σαλαφράγκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι συνεισηγητή ο κύριος Φλάκενστάιν και δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα το πρωί, αλλά μου ζήτησε εκ μέρους και των δύο να κάνω την παρουσίαση στους συναδέλφους. Έχουμε 64 τροπολογίες επί της πρότασης της ε, Επιτροπής που έχει ως στόχο να βελτιώσουμε τον μηχανισμό που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες τις οποίες έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων για αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Το ερώτημα είναι αν θα έχουμε ένα εργαλείο. Είναι σημαντικό το εργαλείο αυτό να συνεχίσει να είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε για την προενταξιακή βοήθεια. Έχουμε πολλά κεφάλαια και παρατήματα και πρέπει να σεβαστούμε τον, χρηματοδοτικό, τον κανονισμό για τα χρηματοδοτικά μέσα. Και αυτός ο κανονισμός προβλέπει τη βοήθεια προς χώρες εκείνες οι οποίες πρόκειται να ε, ενταχθούν κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι, ήταν, ότι είναι προσεκτική η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 14 δισεκατομμύρια προτείνει να είναι το ύψος του προϋπολογισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ε, που θα γίνουν για άλλα χρηματοδοτικά μέσα, όπως για παράδειγμα το μέσο για τη γειτονία. Η κατανομή των κονδυλίων θα πρέπει να γίνεται με ισότιμο τρόπο και στο άρθρο 15 προτείνουμε να καταγραφούν ορισμένα κριτήρια τα οποία να προσδιορίζουμε μεγαλύτερη ακρίβεια τι εννοούμε με ισότιμη κατανομή των κονδύλιων. Πρόκειται για χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται και σε άμεση και σε ε, ε, ε, έμεση διαχείριση και έχουν χρηματοδοτηθεί προγράμματα για την βελτίωση των θεσμών, για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ακόμα και για την βελτίωση του ρόλου που παίζει ο τύπος. Ο γενικός στόχος του EPA3 θα είναι να ενισχύσουμε τις πολιτικές και θεσμικές και μεταρρυθμίσεις, καθώς επίσης και τις μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα ή στην οικονομία που χρειάζονται, έτσι ώστε ε, οι χώρες αυτές να ε, έρθουν πιο κοντά στους πολιτικούς και οικονομικούς και κοινωνικούς κανόνες και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και πιο συγκεκριμένοι στόχοι, τους οποίους μπορεί κανείς να βρει στον κανονισμό, δεν θα αναφερθώ τώρα αναλυτικά, αλλά βασίζονται στις βασικές αρχές, όπως για παράδειγμα το σεβασμό του κράτους δικαίου, την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, την οικονομική ανάπτυξη και την ε, κοινωνική ανάπτυξη, τη συνοχή των περιφερειών κτλ. Κάτι ακόμα που αναφέρεται σε αυτόν τον νέο κανονισμό είναι η μεγαλύτερη δημοσιότητα που θα θέλουμε να δώσουμε στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το οποίο σημαίνει ότι το χρηματοδοτικό εργαλείο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για ε, ενέργειες δημοσιότητας, προβολής του τρόπου με τον οποίο βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα απευθύνονται σε πολλά και διάφορα κοινά. Θα ε, υπάρχει επίσης και ένα ε, σύστημα ε, που θα συμπληρώνει τον κανονισμό, ένα πρόγραμμα εργασιών, το οποίο θα, θένει, θα θέτει πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα και σύμφωνα με το άρθρο 3 θα υποβάλλεται αυτό και κάθε χρόνο για, προς ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Για να λύσουμε προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά το παρελθόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να υπάρξει μια πρόβλεψη για να μπορεί να σταματάει είτε πλήρω είτε μερικώ η προενταξιακή βοήθεια προ μια χώρα η οποία διαπιστώνουμε ότι ε, παραβιάζει τι βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση του κράτου δικαίου με πράξη κατεξουσιοδότη. Στο άρθρο 32 υπάρχουν οι αναφορές στην πολιτική γειτονία και τις διεθνείς σχέσεις ε, και πιστεύω ότι ένα σημαντικό στοιχείο αυτού του ε, κανονισμού, του νέου κανονισμού, είναι ότι θα ενισχύσει το ρόλο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν να ξεκινάει η προγραμματική περίοδος τα σχετικά έγγραφα και Επίσης, θεωρούμε ότι όταν γίνεται η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου. Ε, τα συγκεκριμένα κονδύλια θα καταρτίζονται από το Συμβούλιο με βάση το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και ε, αυτός ο κανονισμός θα δημιουργήσει και μια συστηματική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τη Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση αυτών των χρηματοδοτικών ε, μέσων. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να γνωρίζουμε ακριβώ πώ χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά και ποια προγράμματα χρησιμοποιούνται, ε, ε, χρηματοδοτούνται και πώ υλοποιούνται. Θα δημιουργηθεί επίση και μια συγκεκριμένη επιτροπή για το EPA 3 προς βοήθεια της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς αυτό λοιπόν που ζητούμε είναι να διευκρινιστεί ακριβώς τι σημαίνει η ισότιμη κατανομή, να υπάρχει καλύτερη, καλύτερος συντονισμός των προγραμμάτων, να υπάρχει πλήρης εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να υπάρχει πλήρης εμπλοκή επίσης το, της κοινωνίας των πολιτών και να διασφαλιστεί η διαφάνεια οποτεδήποτε υπάρχει χρηματοδότηση ε, άμεσο, άμεσων προγραμμάτων, προγραμμάτων υπό άμεση διαχείριση. Αυτές τις αρχές τις οποίες προωθούμε στο πλαίσιο αυτού του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού του προγράμματος θα έλεγα ότι θα πρέπει να τις προασπίσουμε και σε οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό ε, μέσο υπέρ τη γειτονία κτλ. θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει μια συνεκτικότητα σε αυτόν τον τομέα, να, να ενισχύσει την εξωτερική διάσταση τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Ευχαριστώ να ακούσω τις απόψεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Ε, εκ μέρου λοιπόν και του κύριου Φλέκενστάιν και ε, εμού. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να παρουσιάσω το προσχέδιο τη εκθεσή μα και ε, ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για να βελτιώσουμε την πρόταση που μας υποβάλλει η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Πριν δώσω τον λόγο στην Κατυπήρη που αντικαθιστά τον Κνούτ Φλέκενστάιν να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών. Υπάρχει μια παράδοση στην πόλη του Αλτενμπουργκ που εκλέγουν ε, τον ε, βασιλιά του Λάχανου εκεί πέρα. Η υψηλότερη πολιτική θέση στην Βόρεια Γερμανία, όλα τα άλλα είναι απλώς οδοντόκρεμες. Ε, καλωσορίζω λοιπόν την αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου υπό την Δήμαρχο. Καλώς ήρθατε. Επανερχόμαστε τώρα σε ζητήματα δημοκρατίας, αφού φύγουμε από τους βασιλιάδες, τον λόγο έχει κάτι πυρί. Δυστυχώς, όπως είπατε, ο Κνούτ Φλέγκενστάιν κόλλιέται, οπότε μου είπε να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλαφράγκα για την εξαιρετική συνεργασία που είχαν και είναι πολύ αισιόδοξο για το ότι τα επόμενα βήματα θα γίνουν στο ίδιο πνεύμα συνεργασίας. Θα διαβάσω την δήλωση του κύριου Φλέκενστάιν. Ζητώ την υπομονή σας. Σήμερα συζητάμε την ε, τρίτη εκδοχή του Μηχανισμού Πενταξιακής Βοήθειας ε, ο οποίος παραμένει εξίσου σημαντικός. Πρόκειται για ένα μοναδικό μέσο που στόχο έχει να προετοιμάσει τις ε, χώρες ε, για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει ένα έργο εξωτερικής πολιτικής, αλλά έχει και μια σημαντική εσωτερική διάσταση για το μέλλον όταν οι χώρες αυτές θα ενταχθούν στην Ένωση. Η εμπειρία που, που κερδίζουν είναι πάρα πολύ σημαντική και για τα διάφορα κονδύλια των εσωτερικών μέσων της Ένωσης για τον ε, μηχανισμό υπαριθμών 3 που θα ισχύσει από το 2021 μέχρι το 2027. Ο Κνούτ Φλέκενστάιν τονίζει πέντε προτεραιότητες. Η πρώτη είναι το ότι θα πρέπει να φαίνεται η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με λύπη διαπιστώνουμε στο παρελθόν ότι σε κάποιες χώρες ε, το κοινό δεν γνωρίζει την βοήθεια που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει στρατηγική σημασία για εμάς, καθώς είναι και άλλοι φορείς πλέον πιο δραστήριοι στην περιοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, ιδιαίτερο στην Σερβία, όπου ο λαός θεωρεί ότι η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στην χώρα, παρά το ότι επενδύει πολύ λιγότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση της Κομισιόν δεν προέβλεπε κάποιες απαιτήσει δημοσιότητας. Ανταυτού υπήρχαν κάποιες ε, αναφορές ε, σε διατάξεις άλλων κανονισμών. Σκοπεύουμε λοιπόν να υπάρξουν συγκεκριμένες απαιτήσεις δημοσιότητας στον κανονισμό του μηχανισμού πενταξιακή βοηθείας. Αυτό πρέπει να το διασφαλίσουν οι δικαιούχοι των χρημάτων αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αντιπροσωπείες της δηλαδή. Δεύτερον, θέλουμε μια δίκαιη κατανομή των κονδυλίων. Ο Κνούτ Φλέγκενστάιν παρατήρησε ότι σε πολλές περιπτώσεις ε, τα χρήματα διανεμήθηκαν μέσω της πρωτεύουσα της ε, κάθε χώρας και όχι εκεί όπου χρειαζόταν και μπορούσε να κάνει διαφορά, αλλά σύμφωνα με πολιτικές πελατειακές σχέσεις. Τα, οι κανόνες μας λένε ότι τα χρήματα πρέπει να μεταφέρουν με τρόπο δίκαιο, χωρίς διακρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιφέρειες. Οι πιο περιφερειοποιημένες περιοχές και εθνοτικές ομάδες πρέπει να κερδίσουν περισσότερο από αυτήν την αλλαγή. Το τρίτο, η πολιτική αιρεσιμότητα, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η πρόταση της Κομισιόν τόνισε ήδη το ότι υπάρχει μια αιρεσιμότητα στο σύστημα και την ανάγκη να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις. Κάτι το οποίο στηρίζει ο Κνούτ Φλακενστάιν. Το σχέδιο της έκθεσης αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στο να γίνουν σεβαστές οι αρχές της δημοκρατίας, πλουραλισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Και θα πρέπει με την εισαγωγή των ρητρών που έχουμε να υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής αφαίρεσης μιας χώρας από τον κατάλογο των χωρών που ωφελούνται από τον μηχανισμό. Και θα υπάρξουν κάποιες πράξεις κατεξιοδότηση προς αυτήν την κατεύθυνση θέλουμε να μετράτε η πρόοδος των δικαιούχων και το κατά πόσον ακολουθούν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει και ένα ελάχιστο ποσό δικαιοσύνη στην κατανομή. Τέταρτον, πρέπει να τονίσουμε την κοινωνική διάσταση της πολιτικής διεύρυνσης. Το σχέδιο έκθεση τονίζει περαιτέρω την κοινωνική διάσταση αυτή. Οι στόχοι πρέπει να είναι απτές, μετρήσιμες αλλαγές ε, στην ε, ζωή των ανθρώπων, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής για, για όσους για το, ειδικά για όσους ανησυχούν για το επίπεδο μετανάστευσης από τα Βαλκάνια. Τα δικαιώματα και οι αρχές που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων τελικά θα ισχύσουν και για αυτές τις χώρες. Οπότε λογικό είναι να καλύπτονται και κατά την εφαρμογή του μηχανισμού προτεξιακή βοήθειας. Επίσης ενισχύουμε την ε, διάσταση της ε, λογοδοσίας με συγκεκριμένους δείκτες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτό αφορά και την ισότητα των φίλων και περιθωριοποιημένων ατόμων. Τέλος, πέμπτο και τελευταίο, ο ρόλος του Κοινοβουλίου έχει μεγάλη σημασία για να υπάρχει δημοκρατική εποπτεία. Ο κύριος Σαλαφράνκα ήδη το ανέφερε αυτό. Ο Κνούτ Φλέκενστάιν έχει και κάποιες άλλες ερωτήσεις ε, για την Κομισιόν. Η πρόταση προβλέπει μια μεγάλη αλλαγή στο πώς γίνονται οι αναφορές. Ε, η Κομισιόν έτσι δίνει στον εαυτό της και μεγαλύτερη ευελιξία και τονίζει περαιτέρω την αιρεσιμότητα με λιγότερα κονδύλια τα οποία είναι εγγυημένα ουσιαστικά για κάθε χώρα. Θα ήθελε όμως ο κύριος Φλεγγενστάιν να μάθει πώς θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό στην πράξη και πώς θα υπάρχει απαραίτητη πολιτική εποπτεία. Συμπερασματικά, ο κύριος Φλέγγενστάιν αναμένει την διεύρυνση της συνεργασίας με τον κύριο Φράγκα και με τους σκιώδης των άλλων ομάδων και των άλλων επιτροπών. και ελπίζουμε να πάμε στον τριμερή διάλογο ε, ενωμένοι ως κοινοβούλιο. Να ευχαριστήσω την Κάτι Πύρη. Για αυτήν την δήλωση που έκανε εκ μέρους ε, του κυρίου Φλέκενστάιν σε σχέση με αυτή την έκθεση του κ. Σαφράγκα και τώρα περνάμε στην συζήτηση. Τρει συνάδελφοι, συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο μέχρι στιγμής. Τρένα Ζόφκο, Αντουντέλη, ο κ. Σαφχάουζα. Υπάρχει κάποιο άλλο συνάδελφο. Μόλι πάνω το λόγο οι συνάδελφοι, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντανιέλσον που παρευρίσκεται εδώ μαζί μα, που είναι εδώ στην αίθουσα. καλώ. Θα του δώσουμε λοιπόν το λόγο έτσι ώστε να απαντήσει και σε κάποια ερωτήματα που έθεσε η κυρία Κάτι πήρε εκ μέρου του κυρίου Φλέκενστάιν. Άρα λοιπόν ε, ξεκινάμε τώρα με τον κύριο Τάνο που είναι ο αρμόδιος και ο από την πλευρά του ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές ε, Σαλαφράκα και Φλέκενστάιν ε, και επιχαίρω το γεγονό ότι ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας έχει παραμείνει ξεχωριστός από το ευρύτερο μηχανισμό της γειτονία και ανάπτυξη. Φυσικά οι ε, διάφορες αυτές ε, χώρες ε, προετοιμάζονται για τη μελλοντική του προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να λογίζουν τον εαυτό του ω απλώ ένα μέλο τη ευρύτερη γειτονία ή τη διεθνού συνεργασία. Οπότε, μόλι θα καταλήξουμε σε ό,τι αφορά το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2021 έω 2027, θα ε, εγκριθεί και αυτό ο μηχανισμό προενταξιακή βοήθεια. Βέβαια, αυτό συνοδεύεται και από μεγαλύτερη ορατότητα του εν λόγω μηχανισμού σε αυτέ τι υποψήφιε χώρε. Ω εγώ μόνιμο ε, εισηγητή σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των πιέσεων που ασκεί η Ρωσία στο Κωσυφοπαίδιο προκειμένου να υπάρξει ένα αντιευρωπαϊκό ή ένα αίσθημα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δείχνει ότι είναι ακόμα πιο επίγον το να καταδείξουμε ακριβώς το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις χώρες. Και ελπίζω το Brexit να αποτελέσει μία και μοναδική ε, περίπτωση όπου έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να καταδειχθεί στην πράξη το τι ακριβώς κάνει στην πράξη η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για αυτές τις χώρες και νομίζω πως ήταν καταστροφικό για τη δική μου χώρα το ότι ακριβώς αυτό δεν καταδείχθηκε, δηλαδή το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Από εκεί και μετά τώρα οι ερεσιμότητες ε, θα πρέπει προφανώς ε, να τις εξετάζουμε ε, και βέβαια δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει εδώ σε αυτή την ε, εξετάζοντας τις θεσιμότητες ε, την Τουρκία. Δηλαδή παρά την μακρά ιστορία και την υποψηφιότητα αυτής της χώρας για σειρά ετών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ζήτημα των κοντιλίων στο πλαίσιο του IPA για την Τουρκία. Πρόκειται για κάτι δηλαδή το οποίο δημιουργεί διαχωριστικές γραμμές μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσα, ανάμεσα στα δικά μας τα ίδια κόμματα. Και, και νομίζω πως θέτει και ένα ζήτημα σε σχέση με αυτούς που υποψήφισαν τον Brexit του 2016. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, καλό είναι να υπάρχει ε, μια ε, επικοδομητική, αν θέλετε, εδώ ε, διαφορά απόψεων σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες ε, μελλοντικής ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση. Πάντως, από εκεί και μετά, η αναλογία που γίνεται μέσα στην έκθεση ε, με το άρθρο 7 είναι, δεν είναι τόσο εύστοχη, γιατί οι υποψήφιες χώρες έχουν την υποχρέωση να προσαρμοστούν στο ενωσιακό και εκτιμένο, αλλά δεν υφίστανται τις ίδιες υποχρεώσεις με τα κράτη-μέλη, τα πραγματικά κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε ένα επιταχυμένο χρονοδιάγραμμα για να εφαρμόσουν ε, τις ε, προποθέσει του ενωσιακού κεκτημένου. Ωστόσο, ε, θα πρέπει ναι και αναγνωρίζω την ανάγκη μιας ρήτρα αναστολής τη διαδικασία για, τι για τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν... Ε, προσαρμόζονται στο κεκτημένο και προβαίνουν σε σοβαρέ παραβάσει. Ε, ε, χαιρετίζω λοιπόν αυτή την, την έκθεση και οι τροπολογίε μα θα έχουν κυρίω συμπληρωματικό χαρακτήρα και δεν θα έρθουν σε αντίθεση με τα όσα προτείνουν οι δύο εισηγητέ. Και ελπίζουμε πω το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει ενισχυμένε αρμοδιότητε ελέγχου και εποπτεία αυτού του μηχανισμού. Σε κάθε περίπτωση πάντω εμεί υποστηρίζουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, τον κύριο Τάνοκ. Ο κύριος Σαφχάουζα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε διάφορες παρατηρήσεις σχέση με αυτή την έκθεση και σχέση με τις τροπολογίες φυσικά. Υπάρχει κάτι που με εκπλήσει. Ότι παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει πολλά κράτη στην πολιτική, την εξωτερική, συζητούμε πάντα το ίδιο. Δηλαδή, λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λειτουργήσει στις συγκεκριμένες σημερινές συνθήκες και βεβαίως να εφαρμόζει τις πολιτικές της για την εξωτερική δράση, για την πολιτική ασφάλεια, για την ε, κλιματική αλλαγή. Παρεπιπτόντως να πω ότι εγώ πιστεύω ότι βεβαίως αλλάζει το κλίμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι ανθρωπογενές. Μιλούμε επίσης για το κράτος δικαίου, αλλά εμείς θέλουμε ένα κράτος δικαίου, όχι ένα κράτος δικαστών. Ακούμε επίσης για προγράμματα για τους μετανάστες, την ε, δίωξη εγκληματιών πολέμου, απλώς εμείς δεν έχουμε τον ίδιο ορισμό για το ποιος είναι εγκληματίας πολέμου. Ε, θα έλεγα ότι είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός για ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις ε, δίωξης. Ακούμε επίσης για αιρεσιμότητα, δηλαδή ότι αν δεν ακολουθήσουμε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να σταματήσει χρηματοδότηση. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σεβασμό για τα κράτη-έθνη, αλλά στην πραγματικότητα προσπαθεί να φτιάξει μια αυτοκρατορία, το οποίο οδηγεί σε πολέμους. Και δυστυχώς παρά τις εμπειρίες που έρχονται, που έχουμε αποκτήσει, συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε χώρες και συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, που θέλουν να ενταχθούν σε αυτήν την Ένωση. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup, monsieur. And we now come to... Σας ευχαριστώ πολύ. Ζελένα Ζόβκο τώρα και συνέχεια ακόμα ένα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους ε, για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης, η οποία παρουσιάζει σωστά το τι θα πρέπει να βελτιωθεί ε, στο μέλλον σε σχέση με τα κονδύλια του Μηχανισμού Προενταξιακή Βοήθειας. Εδώ πραγματικά βρίσκεται στο παιχνίδι η πρόσληψη από τον πληθυσμό ε, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και είδαμε για παράδειγμα ε, στη Βοσνία Ριζεγοβίνη το τι συνέβη στις πρόσφατες εκλογές το ότι δηλαδή επενδύθηκαν κονδύλια από τρίτους προκειμένου να επηρεαστεί το αποτέλεσμα και να προωθηθούν συγκεκριμένοι υποψήφοι. Τώρα η Τουρκία εποφελείται από τα κονδύλια του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποίησε κονδύλια δικά τη για να αυξήσει αυξήσει την επιρροή της στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι υπάρχουν δύο μεγάλοι παίκτες εντός εισαγωγικών, δύο μεγάλες χώρες οι οποίες προσπαθούν να, να καταλάβουν το κενό που άφησε η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί εδώ και πολύ καιρό. Και βλέπουμε την επιρροή που αυτό μπορεί να έχει και στην ε, Βοσνία και στην Κροατία η οποία έχει και το, ε, το μεγαλύτερο σύνορο με αυτή τη χώρα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την χρήση αυτών των κονδυλίων του μηχανισμού ε, νομίζω πως θα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων σε μικρές κοινότητες, η ζωή των ανθρώπων σε μειονότητες των διαφορετικών εθνοτήτων και προκειμένου επίσης να υποβοηθηθεί η διασυνοριακή συνεργασία. γιατί ε, το σχέδιο Μάρσαλ ήταν εκείνο το οποίο προώθησε και τη συμφιλίωση μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο ε, Πόλεμο. Άρα λοιπόν θεωρούμε πως αυτός ο μηχανισμός, ο IPA, θα πρέπει να παραμείνει ξεχωριστός και θα πρέπει να αυξηθεί και μάλιστα όχι μόνο κατά 3% αλλά κατά 4% ή 5% γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η ειρηνευτική διαδικασία και συμφιλίωση στα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Πρόεδρος. Αντορντέλ ε, τώρα. Τρει σύντομε παρατηρήσει. Σχεδιάζοντα τον μηχανισμό προενταξιακή βοήθεια επί τη βάση των ε, ταμείων συνοχή, πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Είναι μια πολύ καλή ιδέα γιατί εκπαιδεύει τα μελλοντικά μέλη Τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμαστούν σε θεσμικό νομοθετικό επίπεδο και σε επίπεδο διοίκηση για το πώς θα χειρίζονται τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Δεύτερον, όσον αφορά του συγκεκριμένου στόχου που θέτει η Επιτροπή, ε, με λυπεί το γεγονό ότι δεν αναφέρεται τίποτα για τις εθνικές και εθνοτικέ μειονότητε, Την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας. Παρά το γεγονό ότι όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί θεμελιώδη αξία τη Ένωση που καθορίζεται και στι συνθήκε και στα κριτήρια τη Κοπενχάγη. Τρίτον, όσον αφορά αυτή τη δυνατότητα να αναστέλλεται η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι σε πολλούς κανονισμούς χρηματοδοτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες απευθύνονται στα κράτη-μέλη, υπάρχουν κριτήρια για το κράτος δικαίου. Ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας αφορά σε κράτη τα οποία δεν είναι ακόμα κράτη-μέλη, είναι κράτη τα οποία προετοιμάζουν τους θεσμούς τους, αξιοποιώντας ακριβώς αυτά τα κονδύλια, έτσι ώστε κάποτε να γίνουν μέλη της Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι το πλαίσιο θα πρέπει να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο. Διαφορετικά, ε, ο μηχανισμός αυτός θα υπόκειται σε έναν πολιτικό ε, σε πολιτικές επιλογές ουσιαστικά τις οποίες θα κάνει η Επιτροπή. Τέταρτον, το ζήτημα της δημοσιότητας. Της δημοσιότητας της Ένωσης. Ε, χαίρομαι για το γεγονό ότι αναδεικνύεται στην έκθεση και πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να προωθείται η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις περιοχές. Η πρόταση ε, το ποσοστό το οποίο θα χρειαστεί να δίνεται για τέτοιες δράσεις δημοσιότητες είναι να, η πρότασή μου την οποία υποστηρίζω να αυξηθεί από το 3 στο 4 ή μέχρι και το 5%. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντέλη, δεν βλέπω κάποιον άλλο συνάδελφο να θέλει το λόγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντάνιελσον. Καλώς ορίσατε κιόλας, είναι η πρώτη σας παρουσία στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ μεγαλειότατε. αστείευεται. Ο μιλητή ξεκινώ πρώτα απ' όλα ε, συγχαίροντας τους συντάκτες της έκθεσής σας. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλά, καλογραμμένη. Προσθέτει ε, ζητήματα ε, και με αυτόν τον τρόπο εμπλωτίζει την πρόταση της Επιτροπής. Μας ικανοποιεί το γεγονό ότι δίνεται έμφαση σε μια στρατηγική προσέγγιση. Προσπαθούμε επίσης, ε, και αυτή είναι η φιλοσοφία του μέσου, να είναι εστιασμένο στα αποτελέσματα, δηλαδή να είναι συγκεκριμένο ο στόχος, το αποτέλεσμα το οποίο ζητούμε και να βλέπουμε αν επιτεύχθη επιτόπου. Έτσι ώστε το κράτος μέλος να συγκλίνει προς τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να γίνει μέλος της Ένωσης. Λαμβάνουμε απόψη μας και σημειώνουμε την σημασία που αποδίδεται σε ορισμένα στοιχεία όπως για παράδειγμα η κοινωνικο-οικονομική σύγκληση. Ε, είναι πολύ σημαντική, για παράδειγμα, και η εκπαίδευση. Γενικώ μιλώντας, προκειμένου ένα κράτος να μπορεί να εντεχθεί. Εξίσου σημαντικές είναι οι τοπικές αρχές, η διασυνοριακή συνεργασία, η κοινωνία των πολιτών. Αναφέρω ορισμένα από τα στοιχεία που θεωρούν σημαντικά. Επίσης, η Επιτροπή σημειώνει την παρατήρηση που κάνατε για τις μειονότητες. Είναι σημαντικό το θέμα. Βέβαια σας παραπέμπω στο παράρτημα 2, ε, το οποίο αναφέρει τους διάφορους τομείς στους οποίους μπορεί να υπάρξει ε, τέτοιο πρόγραμμα παρέμβαση. Και ανάμεσα σε αυτούς τους τομείς είναι και οι μειονότητες. Και έρχομαι στο ζήτημα της δημοσιότητας. Πράγματι, ε, συμφωνούμε και εμείς ότι πρέπει να αυξηθεί. Ακούστηκε το ζήτημα με τη δημοσιότητα σε μία από αυτές τις χώρες ε, και σε άλλες χώρες που απολαμβάνουν βοήθεια από αυτόν τον μηχανισμό υπάρχουν προβλήματα δημοσιότητας και νομίζω πρέπει να αναγνωρίσουμε και κάνουμε μια αυτοκριτική, να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά. Ε, θα πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρη η εικόνα της Ένωσης αξιοποιώντας τη σημαία, αξιοποιώντας το, το, το, το, όνομα και ε, ε, να το προωθήσουμε αυτό μέσω των προγραμμάτων. Είναι ξεκάθαρο ποιο χρηματοδότησε το πρόγραμμα. Έρχομαι σε ζητήματα τα οποία μας ανασυχούν. Πρώτα απ' όλα, η πολιτική ε, της διεύρυνσης είναι μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας είναι ο, ο μηχανισμός για να βοηθήσει αυτή την πολιτική, να την υποστηρίξει και να βοηθήσει τις χώρες που θέλουν να εντεχθούν. Γι' αυτό ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας βρίσκεται και λειτουργεί σε ένα ξεχωριστό διαφορετικό πλαίσιο από άλλους μηχανισμούς που αφορούν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη η οποία χειρίζεται τον μηχανισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ουσιώδους σημασίας. Ε, το βλέπουμε αυτό και στις, σε όλες τις νομικές πράξεις. Ανάμεσα σε αυτές και, τον μηχανισμό, και, συγγνώμη, και την νομική πράξη η οποία θεσπίζει τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας. Αυτό πιστεύω θα πρέπει να το διασφαλίσουμε και να το προσέξουμε στις διατυπώσεις της εκθέσής σας. Για το ζήτημα των πράξεων κάτω εξουσιοδότηση. Ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο έρχεται και ξανάρχεται σε πολλές από τις προτάσεις που υποβάλλει η Επιπεροτροπή. Είναι γνωστή η θέση στη μας. Όμως εδώ συνδέεται και με ένα άλλο ζήτημα. Είναι το ζήτημα της διακυβέρνησης το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο σε βάθος. Είναι ξεκάθαρο και φαίνεται και στην έκθεσή σας πολύ ξεκάθαρα ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να βελτιώσουμε τη, διοίκηση, τη διακυβέρνηση αυτού του μηχανισμού. Υπάρχουν διεστάμενες απόψεις για το πώς μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά θα το διαπραγματευτούμε. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορώ να σας πω ότι θεωρούμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερος, πιο ισχυρός, πιο συστηματικός πολιτικός διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, για τη ρήτρα αναστολής. Ακούσαμε επιχειρήματα που εξηγούν γιατί θα μπορούσε να ήταν χρήσιμος μια τέτοια δυνατότητα. Όμως καταλήξαμε στο, στο, στην απόφαση ότι δεν θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει μια τέτοια ρήτρα σε καθέναν από τους μηχανισμούς, σε καθένα από τα εργαλεία ξεχωριστά. Τούτου λεχθέντος πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε εξελίξεις. Και ε, πιστεύω ότι ήδη έχουμε αυτή τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε σε εξελίξεις. Για παράδειγμα η Τουρκία είναι ένα παράδειγμα όπου συνέβη κάτι τέτοιο. Αυτά είναι τα σχόλια που θα είχε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο στάδιο αυτό τη συζήτηση, αλλά βεβαίω θα συνεχίσουμε και προσβλέπουμε στην, ε, στο διάλογο και στη διαπραγμάτευση μαζί στο πλαίσιο του τριμερού διαλόγου. Ευχαριστώ κύριε Ντέμιλσον. Συνάδελφοι, έχετε σχόλια, ερωτήσει. Όχι. Οι συνεισηγητές θέλουν να πούν κάτι. Κύριε Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις που έκαναν, για τις προτάσεις τους, για ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο. Θέλω να πω ότι ο κανονισμός και έτσι απαντώ και στον κύριο Ντάλη, αναφέρει ήδη στις προτεραιότητες ε, που, για τις οποίες, προωθούμε, τις, τις οποίες προωθούμε και ανάμεσα σε αυτές τις προτεραιότητες αναφέρονται και οι μειονότητες. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι εξάλλου ένα από τα κριτήρια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί λοιπόν και αυτός ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας για, την, για τέτοια προγράμματα, για υπέρ των μειονοτήτων. Το άρθρο τριά επίσης αναφέρεται σε διασυνοριακά προγράμματα και αυτά αναφέρονται ως προτεραιότητα. Ε, έτσι απαντώ και στο ζήτημα που θέτει ο κ. Φλακενστάιν. για το πώς θα μπορούσαμε να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για τα διασυνοριακά προγράμματα. Σημείωσα επίσης και την τοποθέτηση του κ. Ντάνιελσον που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να διατηρήσει να έχει έναν θεμελιώδη βασικό ρόλο στη διαχείριση του μηχανισμού. Ωστόσο, θεωρούμε εμείς ότι και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του ε, ε, Κοινοβουλίου θα μπορούσε να συμπληρώνει, αν θέλετε, να, να εμπλέκεται. Επίση, με τι πράξη κάτι εξουσιοδότηση, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει και καλύτερη εμπλοκή και καλύτερο διάλογο και καλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με το παρελθόν. Και θα συνεχίσουμε φυσικά τον επικοδομητικό διάλογο που έχουμε με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα τη Ένωση, έτσι ώστε τελικά αυτό ο μηχανισμό ε, και να ε, υποστηρίζει και να ε, εξυπηρετεί τους βασικούς μας στόχους και να είναι αποτελεσματικός και να υπάρχει πλήρης εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Καλώ τους συναδέλφους να μας υποβάλουν προτάσεις για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον κανονισμό και έχουμε, θα ήθελα να το πω κλείνοντας, και μια εξαιρετική συνεργασία με τον συνεισηγητή, τον κ. Φρέκενστάιν, και είμαι σίγουρο ότι αντίστοιχη καλή συνεργασία θα συνεχίσουμε να έχουμε και με του κοιόδε και με όλου ε, για όλο το, σε όλη τη διάρκεια που απομένει μέχρι να καταλήξουμε στην τελική έκθεση και να καταλήξουμε σε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράγκα. Ε, κάτι πήρε. Θέλω να προσθέσει κάτι, όχι. Τελειώσαμε λοιπόν την πρώτη εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Η ψηφοφορία είναι στις 4 Φεβρουαρίου. Η Προθεσμία για τροπολογίες είναι η 27 Νοεμβρίου, η ψηφοφορία 4 Φεβρουαρίου. 15 λεπτά μπροστά από το πρόγραμμά μας. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 15 έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία. Η συγκεκριά είναι βεβαίως η συνάδελφος η Κάτι πήρη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Οπότε να δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω λίγο γρήγορα τα κυριότερα σημεία. Για όσους δεν διάβασαν την έκθεση, η έκθεση ξεκινάει από την τρέχουσα κατάσταση στην Τουρκία, εστιάζουμε σε τα κεφάλαια 22 και 23. Καλωσορίζουμε την απόφαση άρσης ε, της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που είχε παρατηθεί 7 φορές και σήμαινε πολλέ παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα όμω λυπούμαστε για το ότι η υιοθέτηση νέων νομοθετικών προτάσεων διατηρεί πολλές από τις εξουσίες αυτές που έχουν δοθεί στον πρόεδρο υπό το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, οπότε ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια αλλαγή από τον τερματισμό αυτών. Υπενθυμίζουμε ότι 150.000 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά το πραξικόπημα και από αυτούς 50.000 ακόμα παραμένουν φυλακισμένοι. Επίσης, από την επιβολή της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, πάνω από 152.000 δημόσιοι υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων δάσκαλοι, γιατροί, πανεπιστημιακοί, εισαγγελείς και δικαστές απολύθηκαν. Και όπως φαντάζεστε οι απολύσεις αυτές είχαν ε, προφανή αντίκτυπο στους ενδιαφερόμενους ε, και τις οικογένειές τους ε, και έχουν ένα μόνιμο κοινωνικό και επαγγελματικό στίγμα. Επίσης η έκθεση καταδικάζει τον αυξημένο έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας ε, στην δικαιοσύνη, στις δικαστές και εισαγγελείς εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τα δυσανάλογα και αυθαίρετα μέτρα που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης των ΜΜΕ και την πρόσβαση στην πληροφορία. Επίσης τονίζουμε το ότι μειώνεται ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών όπου ε, δυστυχώς από όταν κατέθεσα το αρχικό σχέδιο έκθεσης είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την σύλληψη 13 πανεπιστημιακών, ένας εκ των οποίων ακόμα κρατείται Συγκεκριμένη ανησυχία επίσης εκφράζεται για την κατάσταση στα νοτιοανατολικά της χώρας όπου έχουμε σοβαρές κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν ερευνήθηκαν πάρα πολλοί αριθμοί δημάρχων και αντιδημάρχων ε, έχουν απολυθεί ή αντικατασταθεί και ε, αντικατασταθεί από διορισμένους δημάρχους Είχαμε τις δημοτικές εκλογές ε, το Μάρτιο του 2017 και θα πρέπει έτσι να επανέλθει η αρχή της άμεσης δημοκρατικής ε, εντολής ε, των ερετών και στα νοτιοανατολικά της χώρας. Για τους συναδέλφους μας, όπως ξέρουμε, δύο συνάδελφοι, δύο από το Τσέχαπέ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και πολλοί από το ΧΑΝΤΕΠΕ κρατούνται ακόμα και πολλοί από αυτούς πέρασαν από τη φυλακή, μεταξύ των οποίων ε, και η Σελαχατίν Τεμιρτάς, όπου το Εδάδα στο Στρασβούργο χτες έβγαλε μία απόφαση και ζητάει να απελευθερωθεί αμέσως από την προφυλάκηση και γνωρίζουμε ότι η Τουρκία ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, πρέπει να συμμορφωθεί. Μια άλλη περίπτωση που αναφέρεται ε, ακούγεται περίεργο να αναφέρουμε με μονομένα άτομα όταν έχουμε 50.000 ε, κρατούμενους αλλά ε, πρόκειται περί ενός συμβόλου Σμάνα Καβαλά τον οποίο έχουμε σήμερα αντίσει και στο παρελθόν επικεφαλής μιας ΜΚΟ χωρίς πολιτική τοποθέτηση που κρατείται εδώ και ένα χρόνο χωρίς ακόμα να το έχει απαγγελθεί κατηγορία. Μετά για το Κοινοβούλιο πέρσι όταν η Επιτροπή της Βενετίας αξιολόγησε τις αλλαγές του συντάγματος ε, για το νέο προεδρικό σύστημα ήταν σαφής. Το σύστημα αυτό δεν έχει επαρκείς δικλίδες ασφαλείας και κινδυνεύει η διάκριση των εξουσιών ε, μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Και εμείς λοιπόν βάλαμε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή. Εάν παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν όσον αφορά τη δικαιοσύνη, η ελευθερία μίμη, ε, κράτος δικαίου, παραμένουν ως έχουν. Και επιπλέον έχουμε το νέο σύνταγμα που εφαρμόζεται χωρίς ε, να λαμβάνεται υπόψη καμία από τις αξιολογήσεις της Επιτροπές της ε, Βενετίας και του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν το μόνο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι να ζητήσουμε την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Εάν ζητήσουμε κάτι τέτοιο, αυτό βεβαίως σχετίζεται και με τα κονδύλια τα προενταξιακά. Όμως, όπως είπαμε και πέρσι, θέλουμε όλα τα κονδύλια του δεύτερου μέσου και του τρίτου να πάνε σε έναν φάκελο τον οποίο θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πάνε στην κοινωνία των πολιτών για, για προσωπικές επαφές, πανεπιστημιακούς διαλόγους, πρόσβαση των φοιτητών στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και πλατφόρμες για τους μουσιογράφους. Επίσης, έχουμε βάλει στο αρχικό σχέδιο έκθεσης ότι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και 10 χρόνια ζητάει το άνοιγμα των κεφαλαίων 22 και 23 μέσα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ ε, γιατί τα μπλοκάρει το Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, τι ακολουθεί λοιπόν. Εμείς ε, στην Ευρώπη όλοι θα ωφεληθούμε από μια δημοκρατική και σταθερή Τουρκία. Ποια μέσα έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας Στην έκθεση λέω ότι πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή μια πόρτα για τον εξυγχρονισμό και αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης που θα πρέπει να πάει χέρι-χέρι με συγκεκριμένες δεσμεύσεις της Τουρκίας για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, αλλά θα είναι και μια ευκαιρία για ένα πολιτικό διάλογο για την κλιματική αλλαγή και τα εργασιακά δικαιώματα. Για τα εργασιακά δικαιώματα συγκεκριμένα αναφέρουμε στην έκθεση τις συνθήκες εργασίας, ε, την κατασκευή του νέου αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, όπου και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κράτους, 38 ε, εργαζόμενοι πέθαναν σε εργατικά ατυχήματα και υπήρξε και διαδήλωση και 31 διαδηλωτές συνελήφθησαν. Η απελευθέρωση της βίζας σε το Κοινοβούλιο πάντα ήταν σαφές ότι βεβαίως πρέπει η Τουρκία να εκπληρώσει τα 72 κριτήρια μεταξύ των οποίων και ο αντιτρομοκρατικός νόμος αλλά εάν τα εκπληρώσει βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει απαλλαγή βίζας. Η σύνδεση λοιπόν της ατζέντα μας με την αναβάθμιση Τη Τελωνιακή Ένωση και τη απελευθέρωση τη ΒΙΖΑ θα δώσει το μήνυμα και στην τουρκική κοινή γνώμη πω ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στόχο την απομόνωση τη χώρα για την μεταναστευτική κρίση να τηρήσουμε τι υποσχέσει μα. Ε, δηλαδή ε, μεγάλη κλίμακα μεταγκατάσταση και μακροπρόθεσμη χρηματική βοήθεια και τέλο το Κυπριακό βεβαίως που γνωρίζω ότι απασχολεί τους συναδέλφους στο Κοινοβούλιο όπου έχουμε επαναλάβει την παλαιότερη θέση μας όπως πάντα κάνουμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Για τους συναδέλφους ε, που ρωτάνε γιατί δεν υπάρχει το χ και το ψ στην έκθεση, ε, η απάντηση είναι γιατί, όπως ξέρετε, η συγγήτρια έχει περιορισμό λέξεων. Προθεσμία τροπολογιών είναι η 11η Δεκεμβρίου. Ελπίζω, όπως και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, να στείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να μην ε, είναι διαφορετικά τα πράγματα επειδή έχουμε χρονιά εκλογών και παρακαλώ τους συναδέλφους όταν ε, υποβάλλουν τροπολογίες όπως λέμε μην βάλουν πάνω τα πάντα σαν σε χριστουγεννιάτικο δέντρο και αναμένω την συνεργασία με τους ε, συναδέλφους στην πέμπτη χρονιά που κάνουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κάτι πήρε. Έχω τώρα πολλούς συναδέλφους τώρα να πάρουν το λόγο. Ε, η Τουρκία πάντοτε προσελκύει το ενδιαφέρον των συναδέλφων και θα κάνω το εξή. Θα δώσω το λόγο στους και συζητητές για τέσσερα λεπτά στον καθένα και μετά θα δούμε από εκεί και μετά όταν θα πάρουν το λόγο στους και συζητητές πόσος χρόνος απομένει για τους υπολείπους ε, συναδέλφους για τον καθένα από αυτούς. Ε, δίνω τώρα το λόγο στη Ρενάτε Ζωμά από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ε, με κοίταξε συνάδελφο πήρε όταν αναφέρθηκε στο ότι δεν θα πρέπει να υποβληθούν τόσε πολλέ τροπολογίε ώστε να γίνει χριστουγεννιάτικο δέντρο αυτή η έκθεση. Πράγματι, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει σύντομη αυτή η έκθεση, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να, να τεθούν μία σειρά από σημαντικά ζητήματα. Και από εκεί και μετά θα υπάρξουν και τροπολογίε και από τη δική μου πλευρά ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ δηλαδή ότι ε, ε, θα πρέπει να προσθεθούν κάποια στοιχεία ακόμα. Γνωρίζουμε όλοι πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πώς έχουν εξελιχθεί από την τελευταία έκθεση του Ιουλίου δηλαδή του 2017. Ε, πραγματικά είναι κατάλληλη χρονική στιγμή, κατάλληλη συγκυρία για να τοποθετηθούμε πάλι επί αυτού του ζήτηματο. και έχει περάσει αρκετό ε, καιρό από, από το τελευταίο ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Οπότε θα πρέπει να είμαστε σαφεί. Και είναι σαφή η ε, συνάδελφο ε, Κατυπήρη στην έκθεσή τη σε σχέση με ορισμένα σημεία, αλλά σε σχέση με κάποια άλλα θα ήθελα να είναι ακόμα πιο σαφή. Σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου, την ελευθερία τη έκφραση, τι σαφεί υποχωρήσει που έχουν γίνει σε, αυτά τα ζητήματα όπως και το ζήτημα της ελευθερίας της θρησκείας ε, είναι ζητήματα που θα πρέπει να τεθούν ε, με ιδιαίτερη έμφαση. Επίσης, ε, συμφωνώ με το σημείο ιδιαίτερα 13 της έκθεσης, δηλαδή την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και να θυμίσω ότι ο πρόσφατα ο Επίτροπος Χαν έδωσε μια συνέντευξη σε μια γερμανική μερίσια εφημερίδα όπου αξίωσε και εκείνο την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Άρα λοιπόν νομίζω πως αυτό το ζήτημα είναι κάτι το μοιραίο, κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί ακόμα και είναι επιφυλακτική η στάση του Συμβουλίου. Θα πρέπει το Κοινοβουλίο να το υπογραμμίσει ότι θα πρέπει να λάβει χώρα η αναστολή. τώρα, υπάρχουν κάποια σημεία ε, τα οποία λείπουν από την έκθεση και τα οποία είχαν αναφερθεί στην προηγούμενη έκθεση. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Κύπρου η παράγραφος 19 δηλαδή της ε, σημερινής έκθεσης ουσιαστικά δεν ε, ε, ακολουθεί τις συστάσεις που είχαμε κάνει στην ε, τελευταία έκθεση. Για παράδειγμα το ε, πρωτόκολλο της Άγκυρας θα πρέπει να αναφερθεί όχι σε μια αιτιολογική σκέψη αλλά μέσα στα σημεία που θέτουμε και επίσης θα πρέπει να θέσουμε και το ζήτημα των οικισμών στο οποίο προβαίνει η Τουρκία στην Κύπρο. Από εκεί και μετά τα επιθετικά μέτρα τα οποία λαμβάνει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι είναι ένα ακόμα σημείο το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε με μεγάλη σαφήνεια. Αλλά νομίζω πως ε, σε σχέση με αυτά τα σημεία ούτως ή άλλως θα υποβληθούν σωρία τροπολογιών. Από εκεί και μετά δεν έχουν αποσαφινιστεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλλως θα υποβληθουν σωρια τροπολογιων απο εκει και μετα δεν εχουν αποσαφιστει τα προβληματα που αντιμετωπιζει η τουρκια με τις γειτονικέ της χώρες. Για παράδειγμα το κάζους Μπέλη με την Ελλάδα ή το ε, ζήτημα που έχει προκύψει με την Αρμενία γνωρίζουμε πως τα πρωτόκολλα για την εξομάλυνση των σχέσεων με την ε, Αρμενία του 2009 δηλαδή δεν έχουν ακόμα κυρωθεί από την τουρκική πλευρά. Και κατά συνέπεια λοιπόν σταμάτησε και η Αρμενία ε, το Μάρτιο τη σχετική διαδικασία και ίσως και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε. Επίση η ελευθερία της θρησκείας ε, είναι κάτι που θα πρέπει να αναφερθούμε σε ό,τι αφορά και το ζήτημα το αναμένουν δηλαδή από τη μία πλευρά έχουν επιστραφεί οι εκκλησίες και τα μοναστήρια ε, τα οποία είχαν κατασχεθεί παρανόμως αλλά μόνο τα κτίρια και όχι ό,τι τα συνόδευε δηλαδή ε, τα σχετικά ε, κτήματα οι σχετικές εκτάσεις και έχουν τώρα περιέθει στη δημόσια, στην ιδιοκτησία του δημοσίου. Και όταν γίνεται μια αγωγή από την πλευρά των ενδιαφερομένων ε, προκειμένου ακριβώς να λάβουν και πάλι την, ε, να περιέχει πάλι στην κατοχή τους ε, το συγκεκριμένο αγρόκτημα, η συγκεκριμένη έκταση, υπάρχει μία σειρά από διαδικασίες οι οποίες τελικά οδηγούν στην κατάσχεση αυτού του αυτή τη έκταση. Και βέβαια, αν το γνωρίζετε τι συμβαίνει, όταν επιστρέφεται ένα μοναστήρι χωρί την έκταση που το αναλογεί, δεν μπορεί να είναι βιώσιμο αυτό το μοναστήρι. Οπότε ε, θεωρούμε πω αυτό αποτελεί μέρο μια στρατηγική εκδίωξη ουσιαστικά αυτών των κοινοτήτων από την πλευρά τη Τουρκία και θα πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Επίση, θα πρέπει να αναφέρουμε επίση και το ζήτημα τη απαγωγή ε, δασκάλων από τρίτε χώρε, για παράδειγμα όπω την Ουκρανία και την Μολδαβία ε, και αλλού. Και και να πω και κάτι πολύ σοβαρά, αγαπητή κυρία Κατυπήρη. Ε, με λυπεί το γεγονό ότι ξεκινάει η πρώτη παράγραφος με αυτό το welcomes, με το ε, ε χαιρετίζει, με το καλωσορίζει. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεκινάμε με τόσο θετική διατύπωση ε, με μια τέτοια έκθεση. Είναι κάπως υπερβολικό αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να, να διατυπωθεί το συγκεκριμένο σημείο. Ε, υπάρχουν μια σειρά από περαιτέρω ε, παράγραφοι στις οποίες θα μπορούσα να προτείνω την αλλαγή κάποιων ε, σημείων. Για παράδειγμα, εγώ δεν θα ανέφερα το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24, στο πλαίσιο δηλαδή της ε, ενταξιάρχης διαπραγμάτευση. Και από εκεί και μετά έχω κάποιες καλέ ιδέε σε σχέση με κάποιες σημαντικέ τροπολογίες. Ευχαριστώ πραγματικά την εισηγήτρια για αυτή την έκθεση. Αντιλαμβάνομαι πως είναι. Ε, έχει συγκεκριμένου περιορισμού σε ό,τι αφορά την, έκθεση, την έκταση τη και νομίζω πω θα συνεργαστούμε πολύ καλά. Ευχαριστώ, ε, λέει ο πρόεδρος ε, για το ECR τώρα, ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια για το πολύ σοβαρό κείμενο. Ε, έχετε αφήσει πολλά πράγματα εκτός. Διάβασα την έκθεση Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει περιθώριο και υπάρχουν οι περιορισμοί για τις λέξεις, αλλά η εξωτερική πολιτική της ε, Τουρκίας ε, έρχεται κάπως σε σύγκρουση και με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτι άλλο, ένα άλλο θέμα, δεδομένη της μεγάλης τουρκικής διασποράς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις που έχει με το τουρκικό κράτος και τις εντάσεις που έχει αυτό στα διάφορα κράτη-μέλη είναι ένα σημείο το οποίο έχει μεγάλη σημασία αν σκεφτούμε τη μεγάλη επίδραση που έχει το Ίδρυμα Αντιγιανέτ στην τουρκική κοινότητα, στην Ολλανδία και σε άλλες ε, χώρες. Επηρεάζει και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το οποίο είπε η κυρία Σόμερ ε, το αντιλαμβάνεστε και αυτό. Έχουμε και εμείς επαφές ε, με τις ε, διάφορες εκκλησίες ε, στην Τουρκία. Και υπήρχαν πάρα πολλές ανησυχίες για την εξέλιξη που υπάρχει στην τουρκική κοινωνία. Γιατί βεβαίως το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι σε τι είδου ε, καθεστώς ε, μετατρέπεται η Τουρκία επί Ερντογάν. Γιατί αυτά τα οποία βλέπουμε είναι τα συμπτώματα και θα πρέπει να αντιληφθούμε άρα ποια είναι η φύση της ε, κατάστασης. Και υπάρχουν ε, διάφοροι οι οποίοι έχουν πει ότι η Τουρκία πηγαίνει προς ε, μια κατεύθυνση του να καταστεί ένας ε, εκπρόσωπος του Ισλαμικού κόσμου και βλέπουμε ε, ξαφνικά για την υπόθεση Κασόγγι ακούμε ότι πρόκειται περί ενός αντιφρονούς αλλά τι είδους ε, αντιφρονών ήταν αυτός ο άνθρωπος και βέβαια ε, είναι το εντάσσεται στο γενικότερο ζήτημα των ε, σχέσεων που έχει η Τουρκία με τις άλλες ε, γειτονικέ χώρες και ποιος θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι ο κυρίαρχος Ισλαμικού κόσμου να μην μιλήσω βεβαίω για το μίσος το οποίο επικρατεί κατά του Ισραήλ ε, και το τι σημαίνει αυτό και για τους ε, Τούρκους οι οποίοι δεν εντάσσονται σε όλη αυτή την κατάσταση και ανήκουν στο λεγόμενο κοσμικό στρατόπεδο. Τι θέλει λοιπόν ακριβώς να κάνει με την ε, τουρκική δημοκρατία ο Ερντογάν, πώς πάει προς μια κατεύθυνση Ισλαμικής Δημοκρατίας όπως ε, το Ιράν. Πρέπει λοιπόν να δούμε και εμείς ε, τι σχέσεις ε, θέλουμε να έχουμε. Λοιπόν, αναμένω την επικοδομητική συνεργασία μαζί σας, όπως είχαμε και στο παρελθόν και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βέλτα. Επόμενος ομιλητής και πάλι από τις χώρες για την άλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Σχάκη. Ε, δεν θα πω πολλά, η κυρία Κατυπήρη έχει κάνει καλή δουλειά στην έκθεσή της, ε, δείχνει και πάλι και ελπίζω να συνεχίσουμε στον τόνο της συγγήτριας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αρχές ε, και είναι σαφές όταν μιλάμε για τη σχέση μας με την Τουρκία και λυπούμε ε, που μπορώ να πω ότι εμείς είμαστε το μόνο θεσμικό όργανο της Ένωσης ε, που το κάνει αυτό. Χαίρομαι που το πρώτο θέμα της κάτι είναι το κράτος δικαίου, είτε μιλάμε για τις συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που είναι φυλακέ, όπως ο Σμάν Καβαλά, είτε όταν αναφέρεται στα συστηματικά προβλήματα που υπάρχουν με την διάβρωση του κράτους δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, τις ε, δημοκρατικές αυτές αρχές που έχουν κέρια σημασία Επίσης το ότι γίνεται στο διαδίκτυο, η διαδικασία, η κατάσταση των μειονοτήτων, ΛΟΑΤΚΙ, γυναικόπαιδα και τα λοιπά. Και βεβαίως πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας από αυτό και τις σχετικές συνέπειες. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να παραμείνει ανοιχτή η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό έχει ζωτική σημασία, δεν μπορούμε να δεχτούμε απλά μία σχέση εμπορικών συναλλαγών ως εναλλακτικό της ένταξης. Αυτό είναι λάθος. Πάντα πρέπει να έχουμε πρώτες τις αξίες μας και θα επιμείνουμε ε, σε αυτό. Βεβαίως έχουμε δει την εναλλακτική με την κοινική αυτή συμφωνία για το μεταναστευτικό. Πρέπει όμως να αναζητήσουμε καλές λύσεις του λεχθέντος για τους πρόσφυγες που αναζητούν καταφύγιο στην Τουρκία γιατί είναι μεγάλη αριθμή αλλά και οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικέ. και είναι ευθύνη μας να φροντίσουμε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν καλή μεταχείριση και προβλήματα όπως η παιδική εργασία, η σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλα προβλήματα ε, θα αντιμετωπιστούν. Θα αναφερθώ τέλος σε μια επίσκεψη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, στην οποία ήμουν εγώ επικεφαλής. Ε, συναντηθήκαμε με τρεις υπουργούς και όλοι μας μετέφεραν αυτό το οποίο διαβάζαμε και στον τύπο, ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας ενδιαφέρεται για τη βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ ότι είναι καλό το ότι είμαστε σαφείς, ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα λόγια, αλλά οι πράξεις που θα μας πείσουν ότι υπάρχει επικοδομητική νοοτροπία, γιατί υπάρχει τέτοια διάβρωση ώστε ξεκινάμε από πολύ χαμηλό σημείο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη. Και θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε άτομα στην κυβέρνηση. Αυτό περιλαμβάνει και την εισηγήτρια και πραγματικά ελπίζω να μην δούμε τέτοιες δηλώσεις όπως το παρελθόν για την έκθεση που την λένε άκυρη και αυτά τα πράγματα δεν οικοδομούν την εμπιστοσύνη και αν θέλει κάτι τέτοιο η τουρκική κυβέρνηση καλά θα κάνει να αλλάξει τόνο. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην κυρία Βαλέρο από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ. Περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας. συζητούμε εδώ και την έκθεση επί μιας έκθεσης την οποία έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θεωρώ ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι θετικό το γεγονό ότι παρουσιάζεται τώρα και συζητούμε το ζήτημα. Δεν έχει καμία ευθύνη η συγγήτρια, αλλά υπάρχει υπάρξει μια καθυστέρηση. Δηλαδή το 2017 ε, είχαμε ήδη το ΑΦΡΙΜ και θα έπρεπε να είχαμε αναφερθεί σε αυτό. Έχει μια τεράστια συμβολική σημασία. Το λέω αυτό γιατί δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε αυτά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 2017, επειδή απλώς έτσι τεχνικά είναι διατυπωμένη η έκθεση. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2018. Ε, είχαμε της, ε, την δίκη του, ε, είχαμε μάλλον αποστολή παρατηρητών και από το κόμμα μου σε δίκες. Είχαμε τη δυνατότητα να εκφραστούμε εναντίον των παρεμβάσεων στην δικαιοσύνη. και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτών των ε, δικαστικών διαδικασιών θα ήταν διαφορετικό αν δεν είχε υπάρξει τόσο μεγάλη διεθνή κινητοποίηση. Στην περίπτωση του συναδέλφου μας από το αδελφό κόμμα υπήρξε αθώωση, αλλά αμέσως μετά την αθώωση του απαγγέλθηκαν νέες κατηγορίες, ξεκίνησε εκ νέου μια δίωξη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μην σταματήσουμε να δίνουμε ε, την προσοχή μας να φωτίζουμε την κατάσταση στην Τουρκία. Ε, και για να συμβεί αυτό πρέπει να μπορούμε να επισκεπτόμαστε και να έχουμε μια ίδια αντίληψη της κατάστασης επιτόπου. Εγώ είχα την ευκαιρία να, ε, την, να επισκεφτώ περιοχές που επλήγησαν από τον πόλεμο και αντιλαμβανόμαστε ότι στην πραγματικότητα δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα, ότι παραμένουν όπως ήταν και παλιά, όπως παραμένουν στάσιμα. Και το ε, σημαντικό είναι να μην ε, τα παραγνωρίσουμε όλα αυτά για λόγους οικονομικών συμφερόντων. Συνεχίζουν να υπάρχουν περιοχές τις οποίες έχει πλήξει ο πόλεμος, αλλά υπάρχουν και άλλες περιοχές τις οποίες έχουμε κατεδαφίσεις ε, κτηρίων ε, στις, στις περιοχές των Κούρδων προφανώς αναφέρομαι και ε, αυτό καταστρέφει και την πολιτιστική κληρονομιά. Θα υποβάλουμε μια σειρά τροπολογιών για να αναδείξουμε και αυτό το θέμα. Νομίζω ότι το ανέφεραν και συνάδελφοι, ε, θα πρέπει να δούμε εάν θα αποφασίσουμε μια επίσημη αναστολή των διαπραγματεύσεων ένταξης με την ένταξη και τι σημαίνει αυτό και πώς θα καταγραφεί αυτό και στο σημείο 13. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η Τουρκία συνεχίζει να αξιοποιεί τον, μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας γιατί συνεχίζει να είναι υποψήφιο μέλος. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον πιστεύω ότι θα ήταν αντιφατικό ε, ε, να ε, συνεχίσουμε όπως, όπως τώρα. Όσον αφορά την Τελωνιακή Ένωση και αυτήν την, τον εξυγχρονισμό της, συμφωνώ με την κυρία Σάκη. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης εάν δεν υπάρξει αλλαγή της πολιτικής κατεύθυνσης της Τουρκίας προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού. Χρειάζεται να πληρούνται μια σειρά από κριτήρια πριν να έχει νόημα οποιοδήποτε συζήτηση για να συνεχίσουμε έτσι. Και βεβαίω μιλάω για πράξει, όχι για λόγια. Δεν μου αρκεί να ακούω αυτό που θα ήθελε ή αυτό που διακηρύττει ότι θα κάνει κάποια στιγμή η Τουρκία. Ευχαριστώ. Thank you, Valero. Ευχαριστούμε κύριε Βαλέρο. Και τώρα για την QNGL, Δίνω το λόγο στον κύριο Χατζηγεωργίου για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό, ίσως τον τελευταίο χρόνο, η Τουρκία δείχνει κάποια διάθεση στα λόγια επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει επαναλειτουργήσει, μπορώ να το βάλω έτσι, και την ε, Μιχτή Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Επιμένω όμως ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με λόγια γιατί ε, στις πράξεις δεν φαίνεται ότι η Τουρκία είτε κατευθύνεται ουσιαστικά προς τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε προς τον βαθύ εκδημοκρατισμό της χώρας. Θέλω όμως να σταθώ σε ένα ζήτημα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό που είναι η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Προσωπικά νομίζω ότι σήμερα το όνειρο της Τουρκίας για ένταξη έχει αντικατασταθεί από την θέλησή της για αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης. Και νομίζω λοιπόν πως όσοι υποστηρίζουν την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης λέγοντας ταυτόχρονα ότι ε, δεν συζητούν την ένταξη της Τουρκίας πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αντικαθιστούν ε, την, την ένταξη με την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης. Θέλω επίσης να πω ότι όσοι εργαστήκαμε για πάρα πολλά χρόνια προς την κατεύθυνση της ένταξης της Τουρκίας, θεωρώντας ότι αυτή η ένταξη θα μπορούσε να λειτουργήσει ε, βεβαίως προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού της χώρας, αλλά και όσον αφορά εμάς τους Κύπριους και την επίλυση του κυπριακού προβλήματος θεωρώ και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους βέβαια, οφείλουμε να δεχτούμε σήμερα ότι αυτός ο μοχλός έχει, δεν θα πω έχει, έχει εξαϊλωθεί, αλλά έχει μειωθεί πάρα πολύ η, δυνατότητα αυτού του μοχλού να επενεργήσει προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού. Ε, εάν υπάρχει ένας τρόπος, πραγματικά το πιστεύω αυτό, δυστυχώς φάνηκε μέσα από την υποχώρηση του Ερτογάν και την απελευθέρωση του Πάστορα μετά από τις ουσιαστικές πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί εδώ μέσα διαφωνούμε με τον κύριο Τραμπ και εγώ παροσωπικά πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι εκεί απεδείχθηκε πώς και με ποιο τρόπο η Τουρκία μπορεί να κατανοήσει ότι πρέπει να αλλάξει ε, τακτική. Ε, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 28 κράτη-μέλη, με διαφορετικά συμφέροντα κάθε κράτος μέλος, ε, δεν υπάρχει προς, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχει κοινή βούληση προς την κατεύθυνση ουσιαστικής πίεσης ε, στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Σαφάζα για το ΙΕΝΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εάν η Τουρκία δεν ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, ποτέ δεν θα είχαμε συζητήσει την πρώτη αξιακή σχέση. Αυτή η χώρα δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Ευρώπης, παρά μόνο δια της εισβολής σε αυτήν. Ποτέ δεν έχει αποτελέσει μέρος της Ευρώπης ή του πολιτισμού μας. Σήμερα οι συνάδελφοί μου βλέπουν την πραγματικότητα ανακαλύπτουν αυτό που γνωρίζαμε ήδη από την αρχή. Χαίρομαι γι' αυτό που επιτέλους θα τερματίσουμε αυτή την πολιτική την προενταξιακή. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Θα πρέπει να θέσουμε προϋποθέσεις όσον αφορά τους δασμούς και την τελωνιακή ένοξη. Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τι εσωτερικέ τη υποθέσει που τουλάχιστον κανεί θα μπορούσε να πει ότι έχει σχέση με την κυριαρχία, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ούτε τον τρόπο με τον οποίο φέρεται στη διεθνή σκηνή. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε τον Ερντογάν έναν δημοκράτη χριστιανό. Βλέπουμε τι είναι στην πραγματικότητα. Αδελφός μουσουλμάνος. Προσπαθεί να, να, να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να καταστρέψει την Ευρώπη βασικά. Ακούστε τι λέει στο Στρασβούργο, τι λέει στις ομιλίες του στη Γερμανία. Βρισκόμαστε σε πόλεμο, βρισκόμαστε, μια επίθεση ως Ευρώπη και πρέπει να μην του δώσουμε το σκηνή με το οποίο θα μας κρεμάσει. Πρέπει να σταματήσουμε. Τι συζητάμε τώρα για ένταξη, προενταξιακή βοήθεια. Τι νόημα έχει να τα συζητάμε όλα αυτά όταν έχουμε απέναντί μα έναν εχθρό. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι έχουμε έναν εχθρό και να, και να είμαστε ε, αποφασιστικοί. Χαιρετίζω τα θετικά στοιχεία. Σε καμία περίπτωση βέβαια, συμφωνώ και εγώ, πιστεύω και εγώ ότι δεν θα πρέπει να εμπλακούμε στα εσωτερικά της Τουρκίας, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε, πρέπει να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία μας χειρίζεται, μας μεταχειρίζεται, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τους μετανάστες, την Ισλαμοποίηση την οποία υποστηρίζει αυτός ο πρόεδρος, ο οποίος έχει υποστηρίξει τους Ισλαμιστές, ο οποίος έχει υποστηρίξει τους αδελφούς μουσουλμάνους. Όλα αυτά πρέπει να τα πούμε με τρόπο ξεκάθαρο και παρεπιπτόντως για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία εξωτερική δράση αποδεικνύουν την πλήρη ανικανότητά τους και την ανικανότητά τους να αντιληφθούν τι συμβαίνει στον κόσμο. σα. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σαφώ. Κύριος Επιτήδιος τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χιλιάδες εργατόρες έχουν δαπανηθεί ούτως ώστε να συντάσσουμε εκθέσεις σχετικά με το τι συμβαίνει στην Τουρκία, τι πρέπει να κάνει η Τουρκία για να μπορέσει να γίνει μέλο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και το αποτέλεσμα είναι ένα τεράστιο μηδενικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι ο ηγετικό κύκλο τη ε, Ευρωπαϊκή Ενώσεως αντιμετωπίζει το θέμα τη Τουρκία με μεγάλη υποκρισία. Γνωρίζει ότι η Τουρκία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό τη. Γνωρίζει ότι χρησιμοποιεί τη βία είτε απροκάλυπτα είτε και καλυμμένα στη σχέση της με τις ε, υπόλοιπες χώρες. Γνωρίζει ότι απειλεί την Ελλάδα, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και παρόλα αυτά ε, θέλει να δίνει χρήματα και εξακολουθεί να δίνει χρήματα στην Τουρκία, ανέχεται τους εκβιασμούς της Τουρκίας και εμένει στο να την εντάξει με κάθε τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι η Τουρκία μόνο ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι κατά τα λοιπά συζητούμε για αναμόρφωση της ε, τελωνιακής ενώσεως, να καταργήσουμε τους περιορισμούς για την έκδοση βίζας και το κυριότερο, το πιο ουτοπικό, ότι θα δίνουμε χρήματα στην Τουρκία και αυτά θα πηγαίνουν στην κοινωνία των εθνών. Μα η Τουρκία είναι μια δικτατορική χώρα υπό δημοκρατικό μανδύα. Ποιος πιστεύει ότι τα χρήματα τα οποία θα δοθούν για τους πολίτες της Τουρκίας θα καταλήξουν σε αυτούς και θα τα εφαρπάσει ο Ερντογάν. Για όλα αυτά θεωρώ ότι η απειλή για διακοπή των συζητήσεων για την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Επιτιδία. Θα δώσω το λόγο τώρα για τέσσερα λεπτά στην αντιπρόεδρο, στον κύριο Κύρκο μάλλον, ως αντιπρόεδρο της ε, κοινή ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στην Τουρκία. Να ευχαριστήσω τη συνάδελφο την κυρία Πύρη για την πραγματικά βαθιά δουλειά που έκανε σε αυτό το ραπόρτ και να συμφωνήσω απόλυτα μαζί της επίσης ότι τα μέτρα τα οποία δηλώνει η Τουρκία ότι παίρνει μετά το πραξικόπημα είναι πολύ λίγα και πολύ αργά. Και κινούνται πάρα πολύ αργά, τόσο που δεν ξέρουμε αν κινούνται. Εκεί που θα διαφωνήσω είναι στα συμπεράσματα. Η ενταξιακή πορεία, οι διαπραγματεύσει με μάλλον με μια χώρα, είναι ένας τρόπος που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να καθορίσει την εξέλιξη των σχέσεων. Η αναστολή αυτής της πορείας λοιπόν αφαιρεί από το μέρος μας, από τη μεριά μας, ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήσαμε και θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Χατζηγεωργίου, χωρίς μεγάλη αποτελεσματικότητα επί χρόνια, αλλά παραμένει ένα εργαλείο. Και η αναστολή δίνει το μήνυμα και στον τουρκικό λαό ότι η Ευρώπη πια απαγκιστρώνεται καθαρά από τις σχέσεις γιατί να μιλάμε παράλληλα για την, την, τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης, ενώ δεν τον κάναμε, παρά τις δυνατότητες που υπήρξαν από την Κομισιόν, να τον συζητάμε τώρα, αφού δώσουμε το μήνυμα και στην τουρκική κοινωνία, ότι απαγκιστρωνόμαστε από το εργαλείο του εκδημοκρατισμού, πιστεύω πως είναι απλώς για να μην κόψουμε όλα όλες τις γέφυρες, αλλά στην ουσία είναι αναποτελεσματική και ανούσια. Έχει ενδιαφέρον επίσης ότι οι κυβερνήσεις, από ό,τι γνωρίζω, και της Ελλάδας και της Κύπρου, είναι αντίθετες στην αναστολή των διαπραγματεύσεων. Όπως επίσης αντίθετες είναι οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκπρόσωποι των Τούρκων πολιτών, δημοσιογράφοι, πολιτικά κόμματα, όλος ο κόσμος στην Τουρκία με τον οποίο τόσο καιρό διαμορφώσαμε μια σχέση συνεργασίας που δεν είναι η κυβέρνηση φυσικά και όλοι αυτοί μας λένε με μία φωνή μην διακόψετε, μην αναστείλετε τις διαπραγματεύσεις διότι μας ξεπουλάτε. Αυτά πρέπει να τα πάρουμε λοιπόν υπόψη και να δούμε, να κρίνουμε με καθαρό μυαλό ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας στους ψηφοφόρους μας, έρχεται και εκλογικός χρόνος, ποιε είναι οι υποχρεώσει μα στο μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία, ποιε είναι οι υποχρεώσει μα στι γειτονικέ τη Τουρκία χώρε που σηκώσανε το μεγάλο βάρο του προσφυγικού, για το οποίο βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητάει πολλέ φορέ μάταια συμμάχου στη Λιβύη, αλλά ξεχνάμε ότι η Τουρκία και η συμφωνία που κάναμε με την Τουρκία ήταν αυτή που έδωσε στα ανατολικά τουλάχιστον τον περιορισμό του 97% και πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει αν το μήνυμα προς την Τουρκία είναι έχουμε όλες τις πόρτες κλειστές. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συνυπολογίσουμε και εγώ θα προτιμούσα να αφήναμε το de facto πάγωμα των σχέσεων και να μην προχωρούσαμε σε μια ενέργεια η οποία θα εκλειφθεί ως επιθετική από την πλευρά της Τουρκίας. γιατί δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. So, thank you. Σας ευχαριστώ. Α, πήραν τον λόγο οι συνάδελφοι που είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του ω και οι Τώρα περνάω στου υπολείπου συναδέλφου. Δέκα συνάδελφοι ζήτησαν τον λόγο. Και παρότι ξεκινήσαμε αυτό το σημείο τη μέρης σας 20 λεπτά νωρίτερα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε θα δώσω δύο λεπτά στον καθένα από εσά και θα πρέπει να είμαι αυστηρό. Ο κύριο Κούκα πρώτο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την εκτίμησή μου απέναντι στην εισηγήτρια κυρία Κάτι Πύρη ε, για, την, ε, για το ενδιαφέρον που δείχνει για αυτές τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Τουρκίας και επίσης θα ήθελα να την ευχαριστήσω για τη ρεαλιστική της έκθεση. φαντάζομαι ότι δεν ήταν εύκολο να τη συντάξει λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία. Αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση. Ε, θεωρώ πραγματικά και λυπούμε για το γεγονός πως αυτή η έκθεση αποτελεί μια έκθεση που τεκμεριώνει μια επιδείνωση, μια αναχώρηση της υποχώρησης της Τουρκίας σε ό,τι αφορά ε, το κράτος δικαίου αλλά και της θεμελιώδης ελευθερίας. Οι παράγραφοι 4, 4, 5, 6 και 14 είναι πολύ εμφατικέ ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με ε, τη δικαστική εξουσία και τις σχετικές ελευθερίες ε, τηρώντας μια επικριτική στάση, παρόλα αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να αναζητεί ε, τρόπους για να συνεχίσει την επικοινωνία με ε, τους ε, κοινοβουλευτικούς ε, ομολόγους μας, είτε μέσω της σχετικής επιτροπής, είτε μέσω διμερών επαφών σε, σε όλο το πολιτικό φάσμα, έτσι ώστε να διατηρήσουμε τις σχέσεις με τα τμήματα εκείνα της Τουρκίας τα οποία νιώθουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ε, υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε όπως η ε, κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση και η ασφάλεια. Προφανώς αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον η Άγκυρα κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένα θετικό ε, σημείο θα ήταν η εφαρμογή των συστάσεων τη επιτροπή τη Βενετίας σε ό,τι αφορά τι συνταγματικέ τροποποίησει. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, ο κύριο Κούκον. Τώρα ο κύριο Μποστινάρο από την πλευρά των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Κάτι Πύρη για την εξαιρετική δουλειά τη. Πρόκειται για μια εξαιρετική, ρεαλιστική έκθεση που είναι αντικειμενική και πραγματικά αξίζει το δικό μας χειροκρότημα. Ε, όμως εγώ θα έπαιρνα όλα τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση, αυτή την ισορροπημένη τοποθέτηση και επίσης θα λάβανα πολύ σοβαρά τα σχόλια που έκανε ο συνάδελφος, ο αξιότιμος συνάδελφος κ. Κύρκος. Γιατί το πρόβλημα που τίθεται είναι τι κάνουμε από εδώ και στο εξή. Και ποιο είναι το μήνυμα που θα πρέπει να μεταβιβάσει, αν θέλετε, το σημερινό κοινοβούλιο στο επόμενο κοινοβούλιο που θα αναλάβει κοντά. Και εδώ θα κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, είναι θεμελιώδους σημασία να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους διάβλους επικοινωνία ανοιχτού με την Τουρκία, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον σε ό,τι αφορά ειδικότερα και τον εξυγχρονισμό ε, της Τελωνιακής Ένωσης. Αναλογιστείτε δηλαδή τη δυνατότητα υιοθέτηση και εφαρμογή ε, μια ε, τέτοια νέα τελωνιακή ένωση. Γιατί αν δεν το κάνουμε θα χάσουμε δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Και το επόμενο κοινοβούλιο θα ξεκινήσει από το 2020 ουσιαστικά να αναζητεί τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας. Και το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ας ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τομείς δηλαδή στους οποίους για ρεαλιστικούς λόγους και όχι για συναισθηματικούς χρειαζόμαστε πραγματικά ο ένας τον άλλον. Και επιτρέψτε μου να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο κύριε Πρόεδρε. Ας μην τεθεί υπό την ομοιρία συγκεκριμένων ε, εθνικών συμφερόντων αυτή η ατζέντα, αυτό το θεματολόγιο συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Θεοχάρου τώρα από την πλευρά του ΙΣΕΑ έχει το λόγο. Πριν, ε, πριν σας ε, δώσω την παρέμβαση μου, θα ήθελα να ενημερώσω το Προεδρείο ότι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες η Τουρκία απειλεί να με συλλάβει ευθύς ως μεταβώ σε 15 μέρες εκεί στα πλαίσια της Μιχτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εκτελώντας ένταλμα σύλληψης το οποίο είχε καταπέσει και από την Ιντερπολ και από την Europol που έχει εκδώσει το Αζερβαϊτζάν για εντελώ ανόητου λόγου. Το Κοινοβούλιο είναι ενήμερο και ζητώ την προστασία του Κοινοβουλίου, διότι εγώ θα πάω στην Τουρκία και ελπίζω να έχω την προστασία του Κοινοβουλίου. Τώρα, όσον αφορά την αναστολή των ενταξιακών, αυτό ήταν η μοιραία κατάληξη μιας αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς, η οποία στρεφόταν όχι μόνο εναντίον των γειτονικών λαών, όπως είναι η Κύπρος, η οποία τελεί υποκατοχή, αλλά και εναντίον των ιδίων των Τούρκων πολιτών. Ξέρετε κάτω από ποιες συνθήκες ζουν οι Τούρκοι πολίτες. Και βεβαίως κάποιοι, όπως είπε ο κύριος Κύρκος, μας ζητάνε να μην σταματήσουμε τις ενταξιακές και είναι σαν να τους ξεπουλάμε. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι τόσα χρόνια ξεπουλάμε ευρωπαϊκούς λαούς όπως είναι ο κυπριακός λαός που ζει την κατοχή, το ξεκλήρισμα, ε, το εθνικό ξεκαθάρισμα. Ε, η Τουρκία έχει εισβάλει στρατιωτικά και στο Ιράκ και στη Συρία και καταδυναστεύει τους λαούς στους οποίους έχει, ε, ε, κατέχει ε, στις περιοχές τις οποίες κατέχει, ενώ ο εκτουρκισμός ε, συνιστά ε, μια βασική διαδικασία την οποία εφαρμόζει σε κάθε περιοχή που βρίσκεται. Όσον αφορά τον Κυπριακό, εμεί για τόσα χρόνια σα λέγαμε ότι δεν είναι δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λύσει τον Κυπριακό, αλλά να θέσει τι αρχέ και τι αξίε επί των οποίων θα πρέπει να εδράζεται η λύση του Κυπριακού. Ορίστε τώρα που η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, που εμεί λέγαμε ότι είναι apartheid, συνιστά μια ορολογιακή βόβα στα θεμέλια τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα βήμα προ τον πλήρη εκτουρκισμό τη ε, Κύπρου. Εμείς ζητάμε ως βάση επίλυσης του Κυπριακού μόνον όλα όσα προβλέπουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρχές και οι αξίες της, το κεκτημένο χωρίς αποκλήσεις και από την Τουρκία να, να τα σεβαστεί όλα αυτά, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να αναγνωριστεί από την Τουρκία και τα κατεχόμενα να επανενσωματωθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Θεοχάρους. Για δύο λεπτά, κύριο Άλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πύρη, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγητρία για την έκθεση η οποία καλύπτει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να ξεκινήσω μιλώντας για τη μεταναστευτική κρίση σωστά επισημαίνει η κυρία Πύρη τη σημαντικό ρόλο που παίζει η Τουρκία στον έλεγχο του μεταναστευτικού και τη φιλοξενία την οποία έχουν δείξει οι Τούρκοι. Ε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται 3 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες στο, στη χώρα τους. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν προβλήματα με γειτονικέ χώρες όπως και η Βουλγαρία. Υπάρχουν εντάσεις στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και του μεγάλου αριθμού προσφύγων. Μιλάμε για συνολικά σχεδόν 4 εκατομμύρια ανθρώπου. Παρά τις, τις διάφορες δυσκολίες, οι εταίροι μα έχουν αποδείξει ότι έχουν, έχουν αποτελέσει σταθερή δύναμη. Θα έρθω τώρα στο ζήτημα της οικονομίας. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ε, χώρες με τις οποίες έχουμε εμπορικές σχέσεις, έχουμε σημαντικές επενδύσεις. Σωστά το επισημαίνει αυτό η κυρία Πύρη. Πηγαίνουμε όμως και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Η ε, Τουρκία έχει συνεχίσει να προσπαθήσει να ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο, παρά το γεγονό ότι αυτό δεν έχει προχωρήσει όσο γρήγορα θα έπρεπε. Θα πρέπει να το λάβουμε όπως μα και αυτό στην αξιολόγηση τη κατάσταση. Και έχουμε στο κύριο, που είναι το εάν θα γίνει η επίσημη αναστολή των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κυπήρη, εάν αποδεχθεί ε, αποδεχθούμε αυτή την πρόταση. Ποιο θα είναι το πλαίσιο με το οποίο θα συνεργαζόμαστε με την Τουρκία. Αναφέρετε στην εκθεσή σας τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης, που συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικός. Όμως ταυτόχρονα λέτε ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη. Πώς όμως θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτά που θέλουμε εάν θεωρείτε ότι ένας διμερής διάλογος με την Τουρκία θα λειτουργήσει ως σενάριο, πώς θα μπορέσουμε να το προωθήσουμε αυτό αν κάψουμε όλες τις γέφυρες. Θεωρώ επίση ότι μια τέτοια αναστολή θα δημιουργήσει προβλήματα στην κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία και θα απομακρύνει του Τούρκου πολίτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν πρέπει να δεχτούμε. Ε, Αντιθέτω, αυτό που θα θέλαμε να, είναι, θα θέλαμε να ήταν, θα ήταν να ενταθεί ο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστούμε κυρία Άλλη ή κυρία Σακοράφα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι η έκθεση της κυρίας Πύρη περιγράφει την τραγική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ε, Τουρκία και όσα όλα δεν πληρεί όσον αφορά την ε, προενταξιακή της ε, πορεία. Και ορθά επισημαίνει την ανάγκη για επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, όπως επίσης και το πάγωμα των προενταξιακών κονδυλίων. Αλλά την ίδια στιγμή που σημειώνει όλα αυτά, την ίδια στιγμή προτείνει την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης σημειώνοντας ότι θα είναι μια πρώτη τάξεω ευκαιρία για δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει και για την ενίσχυση των σχέσεων καλή γειτονία. Αλήθεια, πιστεύει κανένα μέσα σε αυτή την αίθουσα, κύριοι συνάδελφοι, στα σοβαρά, ότι η Τουρκία θα πάψει να δυναμητίζει την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πάψει τι τυχοδιοκτικέ τη διεκδικήσει σε βάρο ελληνικών και κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων, θα κάνει μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου, θα αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία με την αναβάθμιση Τελωνιακής Ένωσης, με δεδομένο ότι μόλις χθες, το, χθες από κοινοβουλευτικά χίλια ακούστηκε ότι αν χρειαστεί θα ξαναγίνει απόβαση στην τουρκική Κύπρο. Και θεωρούμε ότι αυτό θα είναι η ικανή προϋπόθεση η οποία θα αναστρέψει την κατάσταση που περιγράφει το ψήφισμα. Εγώ μια ανάγνωση έχω εδώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι ε, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρώτα και πάνω από όλα το συμφέρον, τα κράτη-μέλη θα κοιτάνε αδιάφορα, θα πουλάνε υποβρύχια και όπλα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταδικάσει την τραγική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Now we... Σας ευχαριστώ. Κύριος Χριστοφόρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε πραγματικά. Είμαι εξ εκείνων που υπερασπίζομαι νυχθημερών τι αρχέ και τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ένωση δικαίου, όπω καθημερινά το διακηρύσουμε, και ότι βρισκόμαστε εδώ γιατί πραγματικά υπερασπιζόμαστε αρχέ και αξίε. Όσον αφορά το θέμα με την Τουρκία, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Τουρκία παραβιάζει καθημερινά και συνθλίβει κάθε αρχή και αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια από την ημέρα έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ουσιαστικά παίρνει τα πάντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνει χωρί κολλήματα προενταξιακή βοήθεια, συνεχίζεται η Ελληνική Ένωση και η Τουρκία τι κάνει. Τι δίνει η Τουρκία. Η Τουρκία πήρε τα πάντα όλα αυτά τα χρόνια χωρί να δώσει τίποτε. Πλήρη ασέβεια προ όλε τι αρχέ και τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σέβεται το πρωτόκολλο τη Άγκυρα που όφιλε να αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και ήθελα εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, να σα πω πώ θα αισθάνεστον αν η δική σα χώρα βρισκόταν κάτω υποκατοχή από την Τουρκία και την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανήκουμε, έδινε προενταξιακή βοήθεια στην Τουρκία και δεν έπαιρνε καμία κύρωση εναντίον τη Τουρκία. Λέμε καθημερινά για πρόσφυγε και ότι η Τουρκία βοήθησε στο προσφύγο. Μα η Τουρκία δημιούργησε 200.000 πρόσφυγε στην Κύπρο και δεν του αφήνει να επιστρέψουν στι αιστείε του. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία ουσιαστικά δημιουργά προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Προκαλεί καθημερινά δεν σέβεται την κυριαρχία των χωρών μελών, δεν σέβεται την κυριαρχία τη αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κύπρου. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριφερόταν αυστηρά για τα θέματα τη Κύπρου απέναντι στην Τουρκία, εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία δεν θα αποτολμούσε να παραβιάζει με τον τρόπο που παραβιάζει και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό τη και δεν θα τορμούσε να συνεχίσει να προκαλεί. Εγώ στηρίζω το πάγωμα τη ενταξιακή βοήθεια τη Τουρκία και να συνδεθεί αυτό το πάγωμα με την πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην υπόθεση τη Κύπρου. Αλλά ταυτόχρονα θέτω ακόμα ένα ζήτημα. Θεωρώ ότι είναι θέμα ηθική τάξη και αρχή. Χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να πουλούν όπλα στην Τουρκία όταν την ίδια τη στιγμή η Τουρκία χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα για επιθετικού σκοπού, χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα στην Κύπρο, χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα για να βρίσκεται στη Μεσόγειο και να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τη Κυπριακή Δημοκρατία και τη Ελλάδα. Πιστεύω ότι το κλειδί για όλα αυτά τα ζητήματα το πάγωμα των κοντιλίων. Εάν και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, εάν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε αναβάθμιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαν να επιβραβεύουμε για μια ακόμη φορά την Τουρκία και η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι αυτή η απαράδεκτη προκλητική χώρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής, τελευταίοι τέσσερις ομιλητές από τους ε, σοσιαλιστές. Πρώτα ο κύριος Παπατάκης. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια μου στην εισηγήτρια για τη σκληρή δουλειά για να καταθέσει αυτό το report. Η έκθεση αυτή απεικονίζει την πραγματικότητα στην Τουρκία, μια πραγματικότητα την οποία κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν θα ήθελε να είναι έτσι. Όλοι θα θέλαμε να είχαμε μια Τουρκία πραγματικά που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτω ώστε να μπορεί να έχει ένα ευρωπαϊκό δρόμο για να φτάσει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η πραγματικότητα όμω είναι εντελώ διαφορετική. Η Τουρκία είναι μια απέραντη φυλακή, κανένα σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με υπεριαλιστικέ διαθέσει προ όλου του γείτονέ τη, συνεχίζει να κατακρατά το 40% του κυπριακού εδάφους, απειλεί καθημερινά την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, που είναι ευρωπαϊκή οικονομική ζώνη. Δεν ανήκει μόνο στην Κύπρο. Και δεν δίνει το δικαίωμα στην Κυπριακή Δημοκρατία για να προχωρήσει απρόσκοπτα για την αξιοποίηση των υδρογοναθράκων, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν και εναλλακτική πηγή ενέργειας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε πώ συμπεριφέρεται και στους ίδιους τους πολίτες της. Σε καμία περίπτωση η αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία δεν θα πρέπει να σημαίνει αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία. Γιατί θα είναι επιβράβευση από την πίσω πόρτα. Η Τουρκία οφείλει να εφαρμόσει το πρωτόκολλο τη Άγκυρα. Η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί τα δικαιώματα των ίδιων των πολιτών τη. Η Τουρκία οφείλει να έχει σχέσει καλέ γειτονίε με όλα τα κράτη που βρίσκονται στην περιοχή για να μπορέσει να έχει αυτή την ευρωπαϊκή πορεία. Εάν προχωρήσουμε σε αναβάθμιση τη Τελωνιακή Ένωση, είτε στην απελευθέρωση των θεωρήσεων χωρίς η Τουρκία να δώσει κάτι, θα, μπούμε, θα συνεχίσουμε τη λογική αντί καρότο και μαστίγιο, τη λογή καρότου, καρότου που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα και αποδεικνύεται παταγωδός αποτυχημένη. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η Τουρκία διολυσταίνει συνεχώς προς μια αυταρχική και αντιευρωπαϊκή πορεία. Η εφαρμογή του νέου συντάγματος που καθιστά τον πρόεδρο Ερντογάν έναν εκλεγμένο σουλτάνο με απόλυτες εξουσίες, δεν μας αφήνει καμία άλλη επιλογή από το να επιμείνουμε στην απόφαση που είχαμε πάρει πέρυσι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την επίσημη δηλαδή διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Δερμητάς παραμένει φυλακισμένος. Μια φυλάκιση που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου έκανε παράνομη και διέταξε την αποφυλάκησή του. Ο αριθμός Τούρκων πολιτών που ζητά πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα αποδεικνύει, έχει πολλαπλασιαστεί, αποδεικνύει ότι η Τουρκία δεν σέβεται το κράτος δικαίου. Ένα από τα βασικά κριτήρια της Κοπενχάγης που είναι βασικό για την ένταξη. Παράλληλη Τουρκία ενισχύει περαιτέρω την επιθετική της πολιτική. Πρόσφατα, Τούρκοι αξιωματούχοι επανέλαβαν την απειλή πολέμου, το κάζους Μπέλη, ενάντια της Ελλάδος. Συνάδελφοι, συνεχίζονται οι παραβιάσεις στα ελληνικά εναέρια ε, και χωρικά ύδατα και βέβαια έχουμε ισχυρές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ και κινήσεις τουρκικών πλοίων. Τα ζητήματα αυτά, όπως βεβαίω και η προστασία των δικαιωμάτων και του καθεστώτος του, οικονομικού, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα διοκτησιακά δικαιώματα και τα θέματα ελληνικής μειονότητας Ήμβρου και Τενέδου είναι σημαντικά θέματα και πιστεύω ότι πρέπει να περιέχονται στην έκθεση. Βεβαίω, η αγαπητή μου, κάτι που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, επισήμανε να μην γίνει χριστουγεννιάτικο δέντρο το report μέσα από τις πολλέ τροπολογίε. Βεβαίω θα επιτρέψει στου Έλληνε συναδέλφου και του Κυπρίου, λόγω ειδικού ενδιαφέροντο, να βάλουμε μερικά στολίδια παραπάνω σε αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε σχέση με του υπόλοιπου συναδέλφου. Σα ευχαριστώ. Είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη, μεγάλο ενδιαφέρον και από τον αριθμό των Ελλήνων συναδέλφων και Κυπρίων συναδέλφων που πήραν το λόγο. Φαίνεται από το πόσο πολύ ακούστηκαν ελληνικά κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Ο κύριος Μαυρίδης. Ελληνικά θα μιλήσω κύριε Πρόεδρε για ακόμα μια φορά. απολογούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στη μετρική μου γλώσσα όπως είχα πει. Η συγγήτρια όντω χειρίζεται ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα και ίσως πολλοί από εμάς δεν θα ήθελαν να ήμασταν στη θέση της. Και όντω αναγνωρίζουμε ότι αυτή η έκθεση καταγράφει γεγονότα τα οποία θέλει τόλμη για να καταγραφούν. Ξεκινάω με τη διαπίστωση όλων αυτών των αριθμών και της πραγματικής κατάστασης που βρίσκεται στην Τουρκία γύρω από τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, τις παραβιάσεις γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πλήρη περιφρόνηση προς τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, αλλά και το ότι η δικαστική εξουσία στην Τουρκία πλέον είναι ένα πολιτικό όργανο στα χέρια του καθεστώτος. Με αυτές τις διαπιστώσεις όμως, θεωρώ ότι αν ήμασταν ειλικρινείς, θα έπρεπε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι ένα απολυταρχικό καθεστώς. Δεν νοείται δημοκρατία με τέτοιου είδους παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας. Δεύτερο, πώς θα ήμασταν σήμερα αν ακολουθούσαμε διαφορετική πολιτική εδώ και χρόνια. Δεν θα το απαντήσω, θα απαντήσω όμως στο μέλλον. Ας κάνουμε μια αρχή από τώρα. Πρώτον, η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκινώντας από την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεύτερο, μου φαίνεται πράγματι πολύ παράδοξο να δίνουμε αγώνα πώς να αντιμετωπίσουμε την ισλαμιστική πολιτική ατζέντα του Ερτογάν στα Δυτικά Βαλκάνια και να μην δίνουμε αγώνα να απαλλακτούμε από την ισλαμιστική ατζέντα του Ερτογάν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο. Τελειώνω αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι μόνο το κράτος δικαίου που πρέπει να προσπιστούμε, αλλά και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα τα οποία πλήττονται και στα Δυτικά Βαλκάνια και στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκουν αντιμέτωπο την Τουρκία. Thank you. And the final... Ευχαριστούμε. Τελευταίος συνάδελφος, ο κύριος Φροντζούλητσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το επόμενο θέμα είχα ζητήσει το λόγο. Καλό αυτό. Θα σας δώσω το λόγο μετά. Ωραία. Μήπως ο κύριος Ποπόφσκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κύριο Φρέλεσον από την Υπηρεσία Εξωτερικής δράση θα ήθελαν να λάβουν το λόγο. κύριο κύριος Ποπόφσκι πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ε, και χαιρετίζουμε αυτή την έκθεση της κυρίας Κάτι Πύρη που προσπαθεί να αποτυπώσει τα βασικά στοιχεία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας με ισορροπημένο τρόπο. Ε, έχουμε συζητήσει επανειλημμένα αυτές τις ε, σχέσεις κατά την σύνταξη αυτών των εκθέσεων και εμείς συμμεριζόμαστε πολλές από τις ανησυχίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση και τις έχουμε εκφράσει και επανειλημμένα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης, του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας, της δικαστικής εξουσίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν η δική σας έκθεση ευθυγραμμίζεται με τα, τις δυτικά μας επορίσματα και στην ε, ε, σχετική μας ανακοίνωση σε ό,τι αφορά τη διεύνηση Ευρωπαϊκής Ενώσης του 2018. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ σε κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις και αναφορές που γίνονται στην έκθεση. Μας, μας ανησυχεί πολύ ε, αυτή η φυλάκηση μεγάλου αριθμού δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών, αλλά ακόμα και μελών του, της Εθνοσύνδεσης όπως του κ. Ντεμιρτάσε. παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο ήταν πολύ σαφές στην αξίωσή του να απελευθερωθεί άμεσα ο κύριος Δημητάς. Επίσης, η συνεχιζόμενη φυλάκιση ε, του κύριου Ξαγόλου, για παράδειγμα, του κυρίου, που φυλακίστηκε την περασμένη εβδομάδα και του κυρίου Οσμάν Καβαλά, καταδεικνύουν ακριβώς ε, το πρόβλημα που υπάρχει και τα προβλήματα και τις πιέσεις που ασκούνται στην ε, κοινωνία των πολιτών, ε, της οποίας ο χώρος συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί σε αυτές τι ανησυχίε που έχουν εκφραστεί από την πλευρά μα σε ό,τι αφορά την έλλειψη ενός συστήματος ελέγχου, δημοκρατικού ελέγχου, ε, ακριβώς ε, μέσω τη μεταρρύθμισης και του προεδρικού συστήματος ε, και επίσης θεωρούμε πως ε, και πω η σχετική έκθεση που θα συνταχθεί από κοινό με το Συμβούλιο τη Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση τη δικαστική εξουσία θα περιλαμβάνει αντίστοιχε παρατηρήσει. Επίση, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία τη φιλία και το γεγονό ότι δεν καταλήξαμε σε μια συμφωνία λόγω του προπολογισμού, θεωρώ πω θα πρέπει να εγγυηθούμε τα κατάλληλα κονδύλια, ούτω ώστε να επιτύχουμε επαναπροσανατολισμό σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου, τι δημοκρατικέ αρχέ και αξίε και ειδικότερα το ρόλο τη κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή, η Τουρκία πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να συμμετάσχει σε προγράμματα τα οποία ενισχύουν την αμοιβαία μα συνεργασία, όπω για παράδειγμα το Erasmus Plus και το Horizon 2020. Όπω γνωρίζετε, όπω ήδη Ήδη έχουμε προσπαθήσει να αυξήσουμε το σχετικό μέρο των σχετικών κοντιλίων, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών και θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτή την ε, πολιτική μέσα στα επόμενα χρόνια. Και επίση έχουμε αναφέρει με πολύ σαφήνεια στου ε, Τούρκου ομολόγου μα ότι υπάρχουν συγκεκριμένε προποθέσει, αλλά χρειαζόμαστε τα απαραίτητα ε, κονδύλια. Οπότε οι περικοπέ προβλέπονται στον προπολογισμό το 2019 δεν θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να προβεί αυτή την αυξημένη υποστήριξη. Να να πούμε ότι η Τουρκία παραμένει ε, ένας από τους πιο σημαντικούς ε, και εγγύς εταίρους μας, οπότε προφανώς είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει μια σταθερή και δημοκρατική Τουρκία ε, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε το διάλογο με αυτή τη χώρα. Δηλαδή να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας σε μια σειρά από τομείς όπως η ενεργεία, οι μεταφορές, και ούτω καθεξής. Αύριο, είπατε, ο εκπρόσωπο ε, και ο επίτροπο Χάν θα μεταβούν στην Τουρκία για την διαξαγωγή ενό ε, διαλόγου υψηλού επίπεδου με την ε, τουρκική κυβέρνηση και θα γίνουν και κλαδικοί διάλογοι με προσώπου δηλαδή διαφορετικών κλάδων έω τα τέλη του χρόνου σε ό,τι αφορά την ενέργεια και από εκεί και μετά αρχέ του επόμενου χρόνου από τον οικονομικό τομέα. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα που μα ενδιαφέρουν όπω ο εξυγχρονισμό τη Θελωνιακή Ένωση που αναφέρεται και μέσα στην έκθεση που σχετίζονται ακριβώς με τις στενές ε, σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Και επίσης ε, ε, θέλουμε να αυξήσουμε τον διάλογό μας, να τον επιτείνουμε σε ό,τι αφορά την συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη Συρία. Επανερχόμενο στο ζήτημα της, του εξυγχρονισμού της Τελωνιακής Ένωσης, να πω ότι θεωρούμε πως είναι προς το αμοιβαίο όφελος, τόσο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Τουρκίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι το Συμβούλιο θέλει να εκινήσει αυτή τη διαδικασία μόνο ε, εφόσον η πολιτική συγκυρία θα το επιτρέψει. Άρα λοιπόν συνοψίζω λέγοντας ότι μια ουσιαστική συνεργασία είναι δυνατή μόνο εφόσον η ε, Τουρκία σταματήσει με την επιδείνωση πολλών ε, καταστάσεων σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε βελτίωση των τιμερών μα σχέσεων. Ευχαριστώ, λέω ο Πρόεδρο, τον κύριο Ποπόφση ο κύριο Φέρεσεν έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κύριε και κύριοι βουλευτές θα είμαι σύντομο. Δεν θέλω να επαναλάβω τα είπε ο κύριο Ποπόφσκι. Η Υπηρεσία εξωτερική δράση συμφωνεί με την άποψη τη Κομισιόν για την κατάσταση στην Τουρκία και όπω είναι σαφέ, από το εξαιρετικό σχέδιο έκθεση, υπάρχουν πολλοί τομεί σοβαρών ανησυχιών για την κατάσταση στην Τουρκία ιδιαίτερα όσον αφορά το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όπως αναφέρθηκε, η Εκπρόσωπος και ο Επίτροπος Χάν θα πάνε σήμερα στην Τουρκία και στις συναντήσεις τους αύριο θα θέσουν αυτά τα ζητήματα και θα θέσουν ζητήματα που είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία και αποτελούν αντικείμενο συνεργασία όπως ζητήματα εξωτερικής πολιτική. Η Τουρκία είναι πολύ σημαντικός γείτονα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στενός εταίρο ε, και σημαντικό παίκτη σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για την Ένωση. Οπότε έχει κρίσιμη σημασία να συνεχίσουμε τον διάλογό μας με την Τουρκία, να κρατήσουμε ανοιχτούς τους διάβλου επικοινωνία, ε, να ξεπεράσουμε τι διαφορέ μα και να προσπαθούμε να βρούμε κοινέ λύσει. Βεβαίω, είναι ουσιαστικό να υπάρξει μια βελτίωση σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η κοινωνία των πολιτών απαιτεί την εμπλοκή μας στην Τουρκία και χρειάζεται και την οικονομική μας στήριξη. Γι' αυτό έχουμε πολύ σοβαρές επιφυλάξεις, όπως και η Κομισιόν, για τις επιπλέον περικοπές που προτείνονται στο προτεξιακό μέσο να πω επίσης ότι παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά την ε, έκθεση όπως ε, εξελίσσεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Πύρη Μπορείτε να συνοψίσετε σε δύο λεπτά. μισή λεπτό. Αν είναι έτσι για τον κύριο Μπρόκ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την συζήτηση αυτή, η οποία είναι διαφορετική από αυτή που είχαμε πριν από πέντε χρόνια και αυτό δεν είναι γιατί άλλαξε η δική μας ιδεολογία, αλλά άλλαξε η κατάσταση στην Τουρκία. Λοιπόν, δεν θα απαντήσω όλες τις ερωτήσεις γιατί δεν γίνεται αυτό σε δύο λεπτά. Να αναφέρω δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι συμφωνώ, δεν είμαι υπέρ μιας σχέσης που θα αφορά μόνο έτσι, εμπορικές συναλλαγές. Οπότε όποιος θεωρεί ότι η πρόταση του να αναζητήσουμε κάποιες ευκαιρίες στην ε, Τελωνιακή Ένωση χωρίς να υπεραστούμε τις αξίες μας. Προφανώς δεν έχει διαβάσει την έκθεση, δεν ήταν αυτό το μήνυμα το οποίο ήθελε να περάσουμε. Τα στους συναδέλφους που έθεσαν ε, το εάν θα πρέπει επισήμως να ανασταλούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις να πω ότι συμφωνώ. Δεν έχω συναντήσει ούτε έναν στην Τουρκία που να μου έχει ζητήσει να ζητήσω την αναστολή των συνομιλίων. Ούτε η κοινωνία των πολιτών, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε συνδικάτα. Τότε πώς βρίσκεται σε αυτήν την έκθεση. Ε, είναι θέμα αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δηλαδή εάν είμαστε σοβαροί και θα πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν συνομιλούμε με μια χώρα για την ένταξη να έχουμε και καθαρές κόκκινες γραμμές. Και αυτές οι κόκκινες γραμμές έχουν ξεπεραστεί. Και έχουμε τελείως διαφορετικές ιδεολογίες στο Κοινοβούλιο και κάποιοι από 10 χρόνια δεν ήθελαν η Τουρκία να ενταχθεί. Εγώ προσωπικά πάντα θεωρούσα ότι η Τουρκία ανήκει στην Ευρώπη, αλλά κρίνω την κυβέρνηση από την πολιτική της. Και έτσι καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα. Και ως τελική παρατήρηση γιατί ξεπέρασα τα δύο λεπτά. Το να μην κάνουμε τίποτα αυτό το οποίο προτείνουν κάποιοι, Α μην το κάνουμε αυτό. Α μην κάνουμε την τελωνιακή ένωση, α μην κάνουμε το άλλο. Ε, πώς θα μας βοηθήσει αυτό και εμάς για μια πιο δημοκρατική και σταθερή Τουρκία και τους δημοκράτες στην ε, Τουρκία. Οπότε να διαπραγματευτούμε την ε, στρατηγική μας, αλλά να μην λέμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Αυτά και αναμένω τι συζητήσεις αυτές. Σας ευχαριστούμε. Πρόθεσμια για τροπολογίες είναι η 11η Σεπτεμβρίου, 11 η ώρα. Και μια που συζητήσαμε το θέμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, θυμηθείτε ότι η έκθεση αυτή αφορά την ενταξιακή διαδικασία της ε, Τουρκίας και τις σχέσεις ε, με την ε, Τουρκία. Μόνο η σχετικές με αυτό το αντικείμενο ε, τροπολογίες θα γίνουν δεκτές ούτε οξυγενειατικό δέντρο ούτε οτιδήποτε άλλο περνάμε στο επόμενο σημείο 16 και 17 το ένα είναι μέσω χρηματοδοτική στήριξη για τη διαχείριση των συνόρων και θεωρήσεων με εισηγητή τον κύριο Κούκαν και το άλλο είναι θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης ε, κύριο Σουβίστησεν και για τα δύο αυτά θέματα ε, εμείς θα ασχοληθούμε μόνο με την εξωτερική διάσταση και η ΛΥΜΠΕ θα δει την εσωτερική. Η πρώτη για τροπολογίες ήταν στις 9 Νοεμβρίου, η ψηφοφορία είναι στις 6 Δεκεμβρίου θα δώσω τον λόγο τώρα στους δύο εισηγητές για να εκφράσουν την άποψή τους. Θα δώσω τον λόγο πρώτα στον κύριο Κούκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, για την... Ε, τις τροπολογίες τους. Να πω δύο λόγια πρώτα για τη δική μου την προσέγγιση. Εγώ στηρίζω την πρόταση της Κομισιόν το σχέδιο έκθεσης προτείνει ελάχιστες διορθώσεις που προβλέπουν ενίσχυση του δημοσιονομικού πλαισίου για αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων. Θεωρώ τον κανονισμό αυτό ως συνεισφορά στη μεταναστευτική πολιτική στο επόμενο ΠΔΠ. Καλωσορίζω τον αυξημένο δημοσιονομικό φάκελο που έχει αυτό το ταμείο και την αυξημένη ευελιξία που θα πρέπει να έχει. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην συνοχή και τις συνέργειες μεταξύ των μέσων αυτών και όλων των άλλων χρηματοδοτικών μέσων στο πεδίο της μετανάστευσης και διαχείρισης των συνόρων, είτε μέσω του μέσου εξωτερικής χρηματοδότησης ή άλλων μέσων με εξωτερική διάσταση, όπως το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης λίγα σχόλια τώρα. Θεωρώ ότι ο οργανισμός αυτός αποτελεί κομμάτι του μεταναστευτικού πλαισίου που θα πρέπει να φροντίζει για την ε, αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων και το υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφαλείας. Όσον αφορά τον ρόλο των κρατών μελών, θεωρώ πως θα πρέπει να έχουν αρκετή ευελιξία Ταυτόχρονα όμως ε, η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών έχει σημασία κλειδί για την ε, σωστή διαχείριση των συνόρων. Συνολικά υπάρχουν 157 τροπολογίες κάποιες από αυτές ζητάνε διαγραφές όπως σταδιακή κατάργηση των hotspot η σχέση με τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα δεν μπορώ να τη στηρίξω. Χρειάζονται συνέργειες μεταξύ των μέσων και με αυτόν τον τρόπο θα τις εγγυηθούμε. Δεν μπορώ επίσης να δεχτώ τα αιτήματα για διαγραφή της στήριξης τρίτων χωρών. Από την άλλη, ευχαρίστως να στηρίξω την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Edward Kukan and... Ευχαριστούμε κύριε Κούκαν. Και τώρα ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζει η Επιτροπή μας το αυξημένο ποσό που θα αποδοθεί σε αυτό το μηχανισμό με τρόπο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της αγοράς πιο αποτελεσματικά. Θέλουμε επίσης να δώσουμε μεγαλύτερη ε, προτεραιότητα στις, ε, στα μέτρα με τα οποία οι χώρες μπορούν να αντιμετωπίσουν την παράτυπη μετανάστευση συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης. Τονίζεται επίσης η σημασία που έχει να δημιουργηθούν σχέσεις, εταιρικές σχέσεις με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να αποθαρρύνουμε την παράνομη, παράτυπη μετανάστευση. Και ανάμεσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα δημιουργίας κέντρων ε, εξέτασης ετοιμάτων ασύλου εκτός Ένωσης. Θα πρέπει επίση να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν την οδηγία για τις επιστροφές και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι αποτελούν πόλους έλξης για την μετανάστευση στην ε, Ευρώπη και θα πρέπει να μην εξυπηρετήσουμε εκείνους που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες και ε, αναφέρεται ότι οποιαδήποτε οντότητα έχει εμπλακεί σε τέτοιου είδους πράξεις δεν θα μπορεί να ε, δεχθεί χρηματοδότηση, να είναι δικαιούχος χρηματοδότησης. Επίσης υποστηρίζουμε ότι η αρχή της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών και το δικαίωμά τους να επιλέγουν εκείνα από τις διαδικασίες ασύλου αφενός και τις διαδικασίες για τους, την ε, επιλογή των μεταναστών που δέχονται στο έδαφος τους αφετέρου, υπερισχύει της αρχής της ε, αλληλεγγύης. Αυτό λέει η έκθεση, την οποία υποστηρίζω και προσβλέπω στη συνεργασία που θα έχουμε με τον εισηγητή. Ευχαριστούμε κύριε Βίστησεν. Δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, Σκιώδης. Πρώτα. Κύριος Μπρόκ και μετά κύριος Κύριε Μπρόκ. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις από την πλευρά του ΕΛΚΑ σε ό,τι αφορά αυτό το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, ένα ταμείο το οποίο χαιρετίζει η δική μου πολιτική ομάδα. Δηλαδή ενώ ε, χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, άκουσα προηγουμένως και τη συζήτηση για την Τουρκία και ε, βλέπουμε ότι έχει υποδεχτεί στο έδαφος της Τουρκία τον τριπλάσιο αριθμό προσφύγων από τη Συρία σε σύγκριση με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια μας βοηθάει με αυτόν τον τρόπο να έχουμε λιγότερους μετανάστες στην Ελλάδα. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ε, στη συζήτηση που κάνουμε ως προς στον τρόπο που θα συνταχθεί και ε, η έκθεση για την Τουρκία. Η πρόταση τώρα της Επιτροπής είναι μια έκθεση που έρχεται στη σωστή χρονική συγκυρία και ε, ανταποκρίνεται στι αυξημένε ανάγκε για την ε, διαχείριση του αυξημένου αριθμού προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο θα ε, διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται στα δικαιώματα εκείνων οι οποίοι χρήζουν ε, διεθνούς προστασία και επίσης ε, προκειμένου να επιστρέφονται εκείνοι που δεν έχουν το δικαίωμα να παραμένουν με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε την ασφαλέστερη διαχείριση των δικών μας ενόρων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Ε, χαιρετίζουμε λοιπόν αυτή την πρόταση της Επιτροπής ε, και θεωρούμε πως ισορροπεί με το σωστό τρόπο ε, το ζήτημα του ασύλου, της νόμιμης μετανάστευσης αλλά και το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης. Θεωρούμε πως είναι καλά αιτιολογημένη και ανταποκρίνεται με σωστό τρόπο στις προκλήσεις στο επίπεδο της μετανάστευσης. Το ΕΛΚ υπογραμμίζει ότι Εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε μια κοινωνία η οποία βασίζεται στι αξίε τη και μπορεί να είναι περήφανη για τα όσα έχει καταφέρει με βάση αυτέ τι αξίε. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, δηλαδή να τα αποκριθούμε ακριβώ και να σταθούμε στο ύψο των αξιών και των υποχρεώσεων. Πάντοτε υπήρξε αλληλέγγυα Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά συνέπεια πρέπει να είναι αλληλέγγυα απέναντι στους λαούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά και την καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτιών της μετανάστευσης. Ε, στο ε, η αντιμετώπιση της πρόθεσης της μετανάστευσης ε, σημαίνει ότι η αλληλέγγυα στάση των κρατών μελών και ο επιμερισμός ε, του σχετικού βάρους θα πρέπει να είναι κάτι που θα υπερισχύσει. Και σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε από την πλευρά του ΕΛΚ που θα υποβληθούν, να πω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την στενή συνεργασία με τις διάφορες χώρε και να συντονίσουμε μεταξύ του τα διάφορα σημεία και μηχανισμούς εξωτερικής συνεργασίας τη Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να, πάντοτε να επιμένουμε και σε ό,τι αφορά την σύναψη συμφωνιών επιστροφών με, τους, ε, με τις χώρες εταίρους μας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την καταπολέμηση ε, των δικτύων λάτρων μετανάστευσης που πραγματικά δημιουργούν πολύ μεγάλο ανθρώπινο πόνο. Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την περαιτέρω συζήτηση και την επικοδομητική συνεργασία με τις υπόλοιπε πολιτικές ομάδες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπρόκ. Ο κύριος Οντζουλίτσα τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί κύριε Πρόεδρε, καταρχήν ως σκιώδης εισηγητής θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο ε, Κούκαν για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Ε, διάβασα τις συστάσεις του σε σχέση με αυτήν την πρόταση του έκθεση της Επιτροπής και θεωρώ πως τροπολογίες 1 ε, και 2 είναι πολύ σωστές και ισορροπημένες. Ωστόσο δεν είμαι σίγουρος ό,τι αφορά την τροπολογία 3 που προτείνει, δηλαδή μια ημερομηνία λήξης ισχύωσης ε, του κανονισμού. Νομίζω πως αυτό ε, υπερβαίνει λίγο τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Ίσως δηλαδή σε σχέση με αυτό το ζήτημα θα έπρεπε να έρθουμε σε περισσότερη επικοινωνία και να συντονιστούμε με τον εισηγητή της ΛΥΜΠΕ κατά την, τις τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ασφαλή ε, σύνορα και η δημιουργία ενός τέτοιου ταμείου ασύλου και μετανάστευση στο πλαίσιο του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου δείχνει να είναι η σωστή κίνηση. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε πως τα κράτη-μέλη εκείνα ε, τα οποία αντιμετωπίζουν τις υψηλότερες πιέσεις σε επίπεδο μεταναστευτικό θα έχουν τις κατάλληλες δυνατότητες να ανταποκριθούν εξ ονόματος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε λοιπόν πως πρόκειται για ένα μηχανισμό αλληλεγγύης και τον υποστηρίζουμε. Ωστόσο ε, πως ε, πραγματικά θα πρέπει να αποτελέσει μια πραγματική υποστήριξη που ανταποκρίνεται ε, στι ανάγκε των κρατών μελών. Και εδώ αναφέρομαι στι τροπολογίε 13 και 15. Δηλαδή, χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία ε, των εξωτερικών μα συνόρων με κάθε τρόπο, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σεβαστούμε ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία δηλαδή θα πρέπει να αποτελούν πάντοτε τμήμα της αποτελεσματικής διαχείρισης των συνόρων. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε ε, την ε, θέσπιση ε, προγραμμάτων εκπαίδευσης ούτως ώστε να διασφαλίζουμε και την τήρηση των θεμελιωδών αξιών. Και εδώ αναφέρομαι ειδικότερα στην τροπολογία 92. Επίσης το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται σε ό,τι αφορά τις δράσεις σε τρίτες χώρες και η ετήσια έκθεση σε ό,τι αφορά τους διάφορους δείκτες ε, επιδόσεων των διαφόρων χωρών θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε τέτοιε εκθέσει και εδώ αναφέρουμε συγκεκριμένα στην τροπολογία 117. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή τη χρήσιμη έκθεση την ΣΥΤΡΕ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος ε, Λόπες έχει τώρα το λόγο, τελευταίο ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ στην <coughs> έκθεση για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Θα έλεγα ότι για την πολιτική μου ομάδα έχουμε μια διαφορετική θέση από τον εισηγητή, γιατί θεωρούμε ότι αυτό που προέχει είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, ο σεβασμός ε, των υποχρεώσεων μας με βάση αυτό και του ανθρωπισμού. Το οποίο σημαίνει ότι καταρχήν δεν μπορούμε να ε, αποδεχτούμε οποιαδήποτε πρόταση, οποιαδήποτε τροπολογία ξεφεύγει από αυτά. Γιατί γιατί αυτό που γίνεται εδώ με την πρόταση είναι να κάνει μια άμεση σύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης ε, των τρίτων χωρών και την, ε, της αναπτυξιακής βοήθειας μάλλον προς τρίτες χώρες και της συνεργασίας τους για ζητήματα μετανάστευσης με την επιστροφέ, επιστροφές. Δηλαδή ουσιαστικά θέτουμε την αναπτυξιακή βοήθεια υπό προϋποθέσεις δικού μας συμφέροντος. Μειώνεται επίσης το ποσοστό του ταμείου το οποίο θα πάει για, προς ε, όφελος του ασύλου και της, μετα, των διαδικασιών ασύλου και μετανάστευσης. Και ουσιαστικά χρησιμοποιούνται αυτοί οι πόροι, οι οποίοι είναι για το άσυλο και τη μετανάστευση, για κάτι άλλο, δηλαδή για την καταπολέμηση της ε, παράνομης μετανάστευσης. Ε, έχουμε δει τι έχει συμφεί, ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά, με μη κυβερνητικέ οργανώσει οι οποίες δραστηριοποιούνται ε, στη, στον τομέα της, καταπο... της, και μιλούμε επίσης και για οργανώσεις οι οποίες μπορεί να έχουν τιμηθεί ή είχαν υπάρξει υποψήφιε για το βραβείο Ζαχάροφ. Τους τελευταίους μήνε έχει επίση συζητηθεί το ζήτημα και ιδιαίτερα το καλοκαίρι για τα κέντρα ασύλου εκτός ένωσης, το ελάχιστο που μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι ε, αμφιλεγόμενο, τι προτείνουμε ως ε, ομάδα. Θα προτείνουμε μια σειρά από τροπολογίες που θα τονίζουν τη σημασία της ένταξης των μεταναστών. Θα αναφερθούμε στο Διεθνές Δίκαιο για το Άσυλο, τις βασικές αρχές για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη, την ισότητα των φύλων, την πλήρη εφαρμογή του διεθνού δικαίου και ιδιαίτερα όσον αφορά το άσυλο, την καταπολέμηση τη εκμετάλλευση και τη βία. πράγματα δηλαδή τα αποτελούν διεθνεί υποχρεώσει της όλων μας όσον αφορά το άσυλο που προκύπτουν από τη συμβάση της Γενέβης και θεωρούμε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι μεταναστευτικές ζωές βοηθώντας στην ε, καλύτερη ανάπτυξη των τρίτων χωρών με εταιρικές σχέσεις, με πολιτικές σχέσεις με αυτές τις χώρες και τέλος θα τονίσουμε τη σημασία που πρέπει να υπάρχει, που πρέπει να δοθεί σε μια ισότιμη κατανομή των βαρών ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι περίπλοκο. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε ακόμα περισσότερα προβλήματα σε ένα ήδη περίπλοκο πρόβλημα και θα πρέπει να προέχει η αρχή της αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τέλο, σε καμία περίπτωση να μην δαιμονοποιούμε εκείνε τι μη κυβερνητικέ οργανώσει οι οποίε σώζουν ζωέ στη θάλασσα. Έτσι θα, προ... θα προ... Και πορευτούμε εμείς, αυτές τις προτάσεις θα κάνουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε πολύ μακριά από την πιθανότητα να συμφωνήσουμε. Όμως αυτό που χρειάζεται είναι μια πρόταση η οποία θα είναι χρήσιμη για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα περίπλοκο με τρόπο που να σέβεται τις αρχές μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία έκθεση για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης για να περάσουμε ξένα και διαφορετικά πολιτικά μηνύματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω κάποιον να ζητάει το λόγο. Έντουαρντ, ναι, εσύ είσαι εδώ ακόμα στην αίθουσα. Θες να κάτι? Όχι. Οπότε, συνάδελφοι, η ψηφοφορία είναι στις 6 Δεκεμβρίου και μπορούμε τώρα να διακόψουμε και να συνεχίσουμε στις 3 η ώρα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γεωργίας, τον κύριο Ζαλκαλιάνη.